Αν έχετε καλοσύνη, καθίστε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδριασή μας. Έχουμε τους ε, φιλοξενούμενους μας μαζί. Έχουμε τη χαρά να χαιρετήσουμε τις προσωπικότητες και τους εμπειρογνώμονες που έχουμε εδώ μαζί μας για αυτή τη δημόσια ακρόαση που διοργανώνεται από κοινού με το φίλο και συνάδελφο Αντώνιο Παντσέρη με θέμα το να ενισχύσουμε τις θέσεις με τις χώρες γειτονίες και ε, να δούμε και το σε τι στάδιο βρίσκονται σχέση με το Μαρόκο. Έχουμε τον κύριο Λανταμπούρο εδώ που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας τον περασμένο Σεπτέμβριο πριν ε, αναλάβει τα νέα σημαντικά του καθήκοντα του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χαίρομαι που μπορώ να υπογραμμίσω αυτό το, τη νέα, το νέο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και έχουν σημασία ακόμα και τα σημειολογικά στοιχεία όσον αυτό το θέμα. Έχουμε τον κύριο Γιουσέφ Αμράνη που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου που διαπραγματεύτηκε και προσωπικά εφαρμόζει αυτό το θέμα για τον ισχυμένο καθεστώς του Μαρόκου και έχουμε τον Ιβάν Μαρτίν που είναι διευθυντής ερευνών του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών και έχει γράψει πρόσφατα ένα άρθρο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Μαρόκου πώς προχωρήσει, έχουν προχωρήσει αυτές οι σχέσεις και τι γίνεται με τον ισχυμένο καθεστώς ε, θα ήθελα να προβώ σε κάποιες εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις για να σχεδιαγραφήσω τους στόχους και το πλαίσιο της ε, σημερινής μας ακροάσεως. Εδώ και καιρό είδαμε κάποια τάση των γειτονικών χωρών να ανταποκρίνονται θετικά και θα έλεγα να ζητούν επιμόνως διμερείς σχέσεις προνομιούχες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι διάφορες πρωτοβουλίες πλησιάσματο θέτε γητνίασης αποκτούν κάποιες ιδιαίτερες αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε σχέσει για τις, χώρε τις χώρες εταίρους Ευρωπαϊκής Ενώσης και όχι μόνο. Αλλά εδώ αυτές οι σχέσεις ε, είναι πραγματικά ένα εργαστήριο που ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πειραματίζεται με νέε συμβατικές ε, συμφωνίες από αυτέ που ήταν στο πλαίσιο της ε, διευρύνσεως και της ε, πολιτικής ε, γυτνιάσεως. Η πρώτη, στην πρώτη, η πρώτη χώρα είναι το Μαρόκο, στην οποία δώσαμε τον ισχυμένο καθεστώς, αναγνωρίσαμε τον ισχυμένο καθεστώς, εν μεταξύ και το Ισραήλ ξεκίνησε αναβάθμιση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία όμως διεκόπη λόγω της συγκρούσεως στην Γάζα και των διαφόρων προβλημάτων που ακολούθησαν και η Αίγυπτος, η Ορδανία και η Ισία με τη σειρά τους υπέβαλαν αίτημα να συσφίξεως των σχέσεων. αναφέρεται η εταιρική σχέση, η ενισχυμένη εταιρική σχέση πολύ συχνά σαν όρος. Ε, θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο να ετοιμαστεί αυτή η σημερινή συνάντηση όσον αφορά τη συζήτηση των σημαντικών εξελίξεων και να δούμε μαζί με τους επιφανείς φιλοξενούμενους μας εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την προώθηση τέτοιων σχέσεων ε, και αν μπορούν να προωθηθούν μέσω των διαφόρων θεσμών της κοινότητας. Και συμμετέχει και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον καθορισμό της φύσεως των σχέσεων με τους γείτονές μας. Έλειπε μέχρι τώρα η αδίποτε μορφή διαβούλευσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Επιλέξαμε το Μαρόκο ε, διότι θεωρήσαμε ότι είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, πλούσιο σε μαθήματα. Θα δώσω το λόγο στους επαΐοντες, ξεκινώντας από εσά, ε, κύριε Λανταμπούρο. Θα ήθελα να περιοριστούν οι παρεμβάσει ή δυνατόν σε ένα δεκάλεπτο για να αφήσουμε επαρκή χρόνο για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχετε το λόγο κύριε Λανταμπούρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, γιατί όπως γνωρίζετε, σήμερα αρχίζει η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, που προβλέπει αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, οι αντιπροσωπείες που μέχρι χθε ήταν αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 130 σε όλο τον κόσμο, μετατρέπονται σήμερα σε αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διευρυμένες αρμοδιότητες ε, σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και θα εκπροσωπούν πλέον με μόνιμο τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, όλους, ε, τους, ε, σε όλες τις χώρες που είναι παρούσα. Και έτσι στο μέλλον καταργεί αυτές τις ε, εκπεριτροπείς εξάμενες προεδρίες που δεν ικανοποιούσαν ε, την προϋπόθεση μιας συνέχειας στην εξωτερική πολιτική. Ήμουν ε, δύο μήνες στο Μαρόκο και θα προσπαθήσω στο σύντομο χρόνο που μου δώσατε να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις και τη δική μου ερμηνεία για αυτό το περίεργο πλάσμα που είναι αυτό το προηγμένο καθεστώς, το advanced status ή το ενισχυμένο καθεστώς. Θα ήθελα καταρχήν να πω με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου για το προηγμένο καθεστώς αντιστοιχεί σε μια οικονομική και πολιτική εξέλιξη του Μαρόκου, κάτι που επέτρεψε τη συντέλεση προόδου που είναι εμφανής και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το σύμφωνο σύνδεσης εφαρμόστηκε με πολύ καλές προϋποθέσεις και συνέβαλε στη βελτίωση της πολιτικής και δημοκρατικής κατάστασης στο Μαρόκο τα τελευταία δεκαετία και δεύτερον εγγενίασε μια σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξυγχρονιστεί το Μαρόκο και να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη. Δηλαδή το πρώτο θέμα όταν μιλούμε για το προηγμένο καθεστώς, αυτό το advanced status, είναι η αναγνώριση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας ε, ισχυρής τάσης και πρόοδου του Μαρόκου σε ό,τι αφορά την οικονομική, δημοκρατική και πολιτική σύγκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, δεν θα είχαμε προηγμένο καθεστώς αν προηγουμένως δεν είχαμε μία αν δεν είχαμε ένα βαθύ, ξεκάθαρο ε, στόχο και μία δεδηλωμένη και απερίφραστη δέσμευση και προσήλωση του Μαρόκου στη σύγκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ίδιο το βασίλειο του Μαρόκου εφάρμοσε μία διπλωματική στρατηγική με στόχο την σύναψη αυτής ε, της συμφωνίας σύνδεσης, του συμφώνου σύνδεσης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχουμε στο Μαρόκο ένα γείτονα, μια γειτονική χώρα που δεσμεύεται οριστικά και απερίφραστα στην προσέγγιση και στη σύγκλησή του προς την Ευρώπη. Κάτι που σημαίνει ανάληψη δέσμευσης για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προκειμένου να προσαρμοστεί στις αξίες, στις αρχές και στους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια σαφής δεδηλωμένη δέσμευση του Μαρόκου Επίσης, η χώρα αυτή δείχνει μια φιλοδοξία εξυγχρονισμού και εφαρμόζει μια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, για την οποία θα μας μιλήσει, φαντάζομαι, πιο διεξοδικά και ο μεγαλύτερη ακρίβεια ο φίλος Ιουσέφ Αμράνη. Η αναγνώριση της συντελεστής σας προόδου και η δέσμευση του Μαρόκου προς τον εξυγχρονισμό κατέληξαν πριν από ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 2008, σε μία συγκεκριμένη δέσμευση και έναν οδικό χάρτη που προβλέπει αυτό το χρονοδιάγραμμα και το δρομολόγιο για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Αυτός ο δικός χάρτης εντάσσεται στην πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένας μηχανισμός σύγκλησης και πραγματοποίησης αυτών των στόχων. Τι λέει λοιπόν αυτός ο δικός χάρτης, τι λέει αυτό το roadmap, τι λέει αυτό το έγγραφο δέσμευσης υπέρ του προηγμένου καθεστώτος. Καταρχήν, ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη πολιτική διαχείριση των σχέσεων με μια διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Γρανάδα το Μάρτιο στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και που θα είναι η πρώτη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βασιλείου του Μαρόκου. Εν συνεχεία θα βελτιωθεί ο πολιτικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, ώστε να μιλούμε πλέον όχι μόνο για διμερεί θέματα, αλλά στον πολιτικό διάλογο να πραγματευτούμε και άλλα θέματα περιφερειακού ή παγκόσμιου ενδιαφέροντος, για τα οποία καλό θα ήταν να, έχουμε κοινή θέση με το Μαρόκο. Η η πολλαπλή πόλη στον κόσμο, οι συνέπειες ε, της ε, περιβαλλοντικής κρίσης ή της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όλα αυτά τα θέματα που είναι σφαιρικά μας υποχρεώνουν ε, να τα εξετάσουμε και στις διμερείς σχέσεις. Το καθεστώς προβλέπει και την σύγκληση προς κάποιους κοινού κανόνες και αρχές που μας επιτρέπουν και μεγαλύτερη ελαστικότητα. Για παράδειγμα, το βασίλειο του Μαρόκου ανέλαβε τη δέσμευση να πλησιάσει προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και προς τις πολιτικές του. Το Συμβούλιο της Ευρώπης γνωρίζετε όλοι ότι έχει εφαρμόσει πολιτικές που τις εστερνίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι μια υπερφρασμένη δήλωση του Συμβουλίου την Ευρώπη του, του, του, Μαρόκου να συγκλίνει προς το Συμβούλιο της Ευρώπης τα θέματα του πολιτικού διαλόγου. Σε αυτό το προηγμένο καθεστώς ε, θέλουμε να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που θα φέρουν το Μαρόκο πιο κοντά στις οικονομικές και κοινωνικές ε, νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή προβλέπουμε κάποια χρονικά ορόσημα που θα φέρουν το Μαρόκο πιο κοντά στην εσωτερική αγορά και θα τα εντάξουν και όλα στην εσωτερική αγορά. Αυτό συνέβη προηγουμένω και με τι χώρε με τι οποίε έχουμε ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Στην περίπτωση του Μαρόκου, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια ενταξιακή προοπτική. Θα ήθελα να ε, αναφέρω ότι αυτή η σύγκληση είναι η οικειοθελής ε, σύγκληση εκ μέρους του Μαρόκου που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένταξη αλλά για να εξεχωρονιστεί εσωτερικά θέλει να εστερνιστεί το κοινοτικό κεκτημένο σε ορισμένους τομείς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει πριν από ένα χρόνο για το προηγούμενο καθεστώ. Τι συνέβη στο μεταξύ. Έχουμε προχωρήσει τον πολιτικό διάλογο και στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Είχαμε πολύ γόνιμη συνεργασία και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αισθητή πρόοδο ό,τι φορά τη σύγκληση με τις πολιτικές του Συμβουλίου της Ευρώπη. Δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις παρόλο που σε θέματα της γεωργίας έχει οριμάσει η κατάσταση για μια συμφωνία, στο θέμα των υπηρεσιών έχουμε ακόμη δρόμο πολύ να διανύσουμε. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη της ε, κανονιστικής σύγκλησης, δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμη σαφώς τη δέσμευση του Μαρόκου για να ενταχθεί σε αυτή την προοπτική της σύγκλησης. Συντάξαμε και ένα έγγραφο με τους ε, μαροκινούς ομολόγους μας προκειμένου να γίνει μια πιο διεξοδική ανάλυση της κατάστασης που δεν έχω τώρα το χρόνο να σας τα παρουσιάσω. Είδαμε τα βήματα που έγιναν προκειμένου να εφαρμοστεί και εμπράκτως αυτή η σύγκληση και εντοπίσαμε και τις α, ε, μελλοντικές προκλήσεις, τις πιο σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις. Και με αυτό θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε τις οικονομικές και εμπορικές διαπραγματεύσεις που εκκρεμούν ώστε μετά την ολοκληρωσή τους να εγγενιάσουμε μια νέα εμπορική και οικονομική συμφωνία πιο βαθιά και πιο φιλόδοξη, ώστε να έχουμε πραγματική σύγκληση των οικονομικών τελεστών και να συμπεριλάβουμε κάποιο τρόπο, να εντάξουμε κάποιο τρόπο το Μαρόκο στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα είναι ο πρώτο στόχο θα δούμε τι θα συμβεί του επόμενους μήνες. Πάντως, η αξιοπιστία του προηγμένου καθεστώτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα που θα επιδείξουμε του επόμενου μήνες να ολοκληρώσουμε τις εκκρεμίε διαπραγματεύσει και να θέσουμε και έναν πιο φιλόδοξο ορίζοντα. Δεύτερη πρόκληση, που αποτελεί ταυτόχρονα και τον πυρήνα ή την πεμπτουσία αυτού του προηγμένου καθεστώτος, είναι το σχέδιο κανονιστικής σύγκλησης. Οι μαροκινοί φίλοι μας θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να προσδιορίσουμε σαφήνεια το επίπεδο των φιλοδοξιών τους σε ό,τι αφορά την κανονιστική σύγκληση. Θα πρέπει να μας πούν από ποιους τομείς θέλουν να ξεκινήσουμε. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ανταγωνισμό, ή κάτι άλλο. Και μαζί να καθορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε την υλοποίηση των στόχων, τις δεσμεύσεις και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Ώστε να καταμετρήσουμε την πρόοδο, την εξέλιξη ή ενδεχομένως και την αποτελμάτωση ή το διέξοδο. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό για να προβούμε σε μια αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση της πρόοδου. Αυτό θα επιδιώξουμε τους επόμενους μήνες. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Απαιτεί βέβαια κολοσιαίο έργο και τεράστια προσπάθεια εκ μέρους της μαροκινής κυβέρνησης και διοίκησης. Πάντως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τους δύο μήνες που είμαι στο Μαρόκο έχω πιστεί ακράδαντα για την ε, ουσιαστική δέσμευση της μαροκινής κυβέρνησης και της μαροκινής διοίκησης για να δοθεί σάρκα και οστά στο προηγμένο καθεστώς, που είναι και φιλόδοξο και περίπλοκο. Αν όμως καταβληθούν αυτές οι τεράστιες προσπάθειες, θα καταφέρουμε να επιφέρουμε μια προστιθέμενη αξία στην ε, Συμφωνία Σύνδεσης. Σήμερα το Μαρόκο είναι η μοναδική χώρα με την οποία έχουμε συνάψει ένα τέτοιο προηγμένο καθεστώς δεν πρόκειται για έναν ιδιάζοντα νομικό κανόνα, αλλά πρόκειται για μια πολιτική δέσμευση που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες και απτές ε, δεσμεύσεις που ενισχύουν το διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό και συσπηρώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο για να αντιμετωπίσουν τις ε, παγκόσμιες ε, κρίσης αλλά και το δράμα του μεσανατολικού ζητήματος. Αν λοιπόν εργαστούμε και εμείς και το Μαρόκο καλά, ιδιαίτερα το Μαρόκο, θα βρεθούμε σε μια καλύτερη γειτονική σχέση που θα μας εξασφαλίσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο. Σας ευχαριστώ κύριε Λανταμπούρου. Ο κύριο Ιωσέφ Ανουράνη, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια ακρόαση που λαμβάνει η χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ακρόαση που για μας, ε, για το Βασίλειο του Μαρόκου, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όπως είπε και ο πρέσβης Λανταμπούρου, οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου έχουν και για την πατρίδα μου στρατηγική σημασία. Το Μαρόκο ανέκαθεν ζητούσε αυτή την ε, έναρξη αυτής της διαδικασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει όλο και μεγαλύτερη σύγκληση μαζί της. Και όπως είπατε, και εσείς κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε ανέκαθεν το Μαρόκο ως προνομιακό εταίρο στην Ευρωμεσογειακή Λεκάνη. Ως εκ τούτου και η σημερινή μου παρουσία εδώ μας γεμίζει με ικανοποίηση και εμάς, αλλά φαντάζομαι και εσάς. Γιατί για το Μαρόκο η σύνδεση με την Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα, προτεραιότητα της κυβέρνησης και μάλιστα όχι μόνο στρατηγική προτεραιότητα, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη υποδειγματικών σχέσεων. Όπως ξέρετε, από τις 13 Οκτωβρίου του 2008, το Μαρόκο γεννίασε ένα νέο στάδιο στη Συμφωνία σύνδεση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που κατέστη δυνατό χάρη στην υιοθέτηση ενός κοινού εγγράφου του οδικού χάρτη που προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των σχέσεων μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των βασικών μας ε, στόχων για όλους τους τομείς που μας ενδιαφέρουν και για όλες τις πτυχές που μας ενδιαφέρουν. Βέβαια, μέσα σε ένα δεκάλεπτο είναι πολύ δύσκολο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα σημαντικότερα ορόσημα αυτής της διαδικασίας που κατέληξαν στην νέα αυτή εταιρική σχέση, να προσδιορίσω τη φύση του, τους στόχους του και τέλος να αναφερθώ στις μελλοντικές μας προοπτικές. Εν συντομία, το βασίλειο του Μαρόκου εργάστηκε ανέκαθεν υπέρ της εμβάθυνσης των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πνεύμα της συνθήκης της Ρώμης. Και αυτό κατέστησε σαφές μέσω μιας εμπορικής συμφωνίας που ήδη υπογράψαμε από το 1969 με την τότε Ευρωπαϊκή και Οικονομική Κοινότητα αλλά είχαμε και μια σφαιρικότερη συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε το 1976. Πάνω από 14 χρόνια μετά την ε, συνθήκη της Βαρκελ... τη διάσκεψη της Βαρκελόνης και πάνω από 9 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σύνδεσης και πάνω από 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ε, της γειτονίας, ήταν φυσιολογικό και απόλυτα αναμενόμενο να επιδιώξουμε μια ευάθυνση των σχέσεών μας και την υιοθέτηση ενός πιο φιλόδοξου και πιο συγκεκριμένου πλαισίου. Έτσι, είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα του υπάρχοντος πλαισίου σύνδεσης. Και όπως είπε και ο Ενέκο Λανταμπούρου, αυτή είναι μια φιλοδοξία, ήταν μια φιλοδοξία του Μαρόκου, αλλά ταυτόχρονα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, Μαρόκο είχε ανέκαθεν εκφράσει τη βούλησή του να, αποτελεί, να αποτελέσει τμήμα μιας όλο και πιο φιλόδοξης και βελτιωμένης διαδικασίας. Και αυτό εξηγείται από τη στρατηγική τοποθέτηση του Μαρόκου, που είναι προνομιακή, βρίσκεται μόνο 14 χιλιόμετρα από την Ευρώπη και έχει πάρα πολλά σημεία που το φέρνουν κοντά στην Ευρώπη. Μάλιστα, το περιβάλλον το επενδυτικό στο Μαρόκο είναι παρόμοιο με αυτό που ισχύει στην Ευρώπη. Η μαροκινή οικονομία εκπληρώνει τα μακροοικονομικά κριτήρια του Μάστριχτ. Είναι μια ισχυρή, εύρωστη και σταθερή οικονομία και έχει μειωμένο έλλειμμα. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που θεσπίστηκε το 2003 και μάλιστα το Μαρόκο ήταν από τις πρώτες χώρες του Νότου που υποστήριξαν αυτή την πολιτική γειτονίας. Η πολιτική αυτή έχει ως βασικές αρχές τη διαφοροποίηση και την ενισχυμένη συνεργασία. Και αυτή ήταν μια πρώτη απάντηση στη φιλοδοξία του Μαρόκου. Με βάση αυτές τις δύο αρχές η χώρα μου κατέβαλε σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που από την αρχή υποστηρίξαμε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Το προηγμένο καθεστώς, όπως έχει αποκρισταλωθεί, αντικατοπτρίζει τη βαθύτατη και στρατηγική φιλοδοξία του Μαρόκου. Γιατί το Μαρόκο χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιζητεί τη συνεργασία μαζί της και τις ενισχυμένες σχέσεις. Αυτό όμως δείχνει και την υποστήριξη που μας έδωσε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις στρατηγικές μας επιλογές. Αλλά αυτό φάνηκε και από τη διαδικασία εξυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού που προώθησε ο βασιλέας του Μαρόκου. Σε ό,τι αφορά το προηγμένο καθεστώς, θα ήθελα να πω ότι για το Μαρόκο, πριν την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων, ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων του Μαρόκου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θελήσαμε μια πολύ συμμετοχική και ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης. Θέλησαμε να βεβαιωθούμε για την υποστήριξη όλων των ε, θεσμικών και πολιτικών φορέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θελήσαμε δηλαδή να εφαρμόσουμε παρόμοια δυναμική με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το έγγραφο που εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008 χαράζει έναν οδικό χάρτη που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δράσεις και σχέδια με έναν ισορροπημένο ρυθμό μεταξύ των τριών διαστάσεων ε, του προηγμένου καθεστώτος που είναι η πολιτική, η οικονομική και η ανθρώπινη διάσταση. Γιατί τώρα αυτό το προηγμένο καθεστώς, το ενισχυμένο καθεστώς. Γιατί το Μαρόκο επέτυχε μία νέα δυναμική και μία νέα συσφίξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και φάνηκε η ανάγκη ενός πιο ενισχυμένου πλαισίου για τις σχέσεις μας. Είχαμε ήδη μια ενδιαφέρουσα εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχαμε στο παρελθόν σε πολλές ειρηνευτικές επιχειρήσεις, όπως την επιχείρηση Αλτέα. Είχαμε συνάψει σημαντικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Συμφωνία Open Sky και Γαλιλαίο. Οπότε ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό να ενταχθούμε σε μια νέα φάση των σχέσεών μας. Ένα χρόνο μετά το 2008, τη σύναψη της Συμφωνίας για το προηγμένο καθεστώς. Τι καταφέραμε. Πιστεύω ότι σε πολιτικό επίπεδο είχαμε σημαντικά επιτεύγματα. Καταρχήν, ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας με την ε, ΚΟΠΣ, την ε, Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, και μάλιστα είχαμε ανταλλαγές για σημαντικά θέματα ασφάλειας με τους εταίρους μας, όπως τις τρομοκρατικέ απειλές στις διόχθες του Ατλαντικού και έχουμε ένα μηχανισμό διαλόγου και συνεργασίας όπου μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς με τη δική μας οπτική γωνία. Και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο και για το Μαρόκο αλλά και για τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μάλιστα είχαμε πολιτικές διαβουλεύσεις και με την Σουηδική Προεδρία. Μάλιστα είχαμε και μια συνεδρίαση παράλληλη με την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ήδη ξεκινήσαμε διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και γενικώ έχουν εγκαινιαστεί πολλές πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος. Έχουμε πια πολύ στενή σχέση και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και γενικώ προχωρούν καλά τα πράγματα στην πολιτική διάσταση. Τώρα, έρχομαι στη δεύτερη οικονομική διάσταση, αλλά προηγουμένω ήθελα να πω δύο λόγια για την κοινοβουλευτική διάσταση. Από αυτή την άποψη θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερη σημασία που δίνει το Μαρόκο στην κοινοβουλευτική διάσταση και στην ανάγκη ενίσχυσης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου. Γι' αυτό και θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να απευθύνω μια έκκληση να συγκεκριμενοποιηθεί το συντομότερο δυνατό αυτό ο διάλογο και να συστηθεί αυτή η μεικτή επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίου του Μαρόκου. Γιατί το Μαροκινό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο και μάλιστα ε, συγκάλεσε και έκτακτη σύνοδο, παρουσία δύο Ευρωπαίων πρεσβευτών, για να ασχοληθεί με το θέμα του προηγμένου καθεστώτος. Γιατί στο Κοινοβούλιο του Μαρόκου τα πολιτικά κόμματα έχουν πολλές προσδοκίες από το προηγμένο καθεστώς και από τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ηγερθεί τεράστιες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την οικονομική διάσταση. Την ανέφερε και ο κύριος Ενεκό Λανταμπούρου. Νομίζω ότι σε οικονομικό επίπεδο το πιο σημαντικό είναι η κανονιστική σύγκληση σε θέματα εσωτερικής αγοράς. Το Μαρόκο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έχει προτεραιότητα αυτή τη σύγκληση. Θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στην εσωτερική αγορά. Και είμαστε διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να προχωρήσουμε στα, στις διαπραγματεύσεις και για την απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών και το δικαίωμα της εγκατάστασης, αλλά και στα γεωργικά θέματα. Μάλιστα, η στρατηγική θέση για την σύναψη μιας νέας συμφωνίας και μια καλύτερη, καλύτερη ενσωμάτωση του Μαρόκου στην εσωτερική αγορά είναι βασική στόχη της χώρας μου. Βέβαια, το φιλόδοξο προηγμένο καθεστώς δείχνει την δέσμευση όλων των κλάδων του Μαρόκου προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους οικονομικούς τελεστές και τους επιχειρηματικούς παράγοντες, ώστε να υποστηρίξουν, να συμμετέχουν και να προωθήσουν τη συμφωνία του προηγμένου καθεστώτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα επιτεύγματα του οικονομικού κεφαλαίου, θα ήθελα να τονίσω την σύγκληση της νομοθεσίας σε θέματα καταπολέμησης παραποίησης, πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή και τη σύσταση του Μαροκινού Γραφείου Προστασίας του Καταναλωτή. Τώρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη διάσταση, έχουμε προσέγγιση θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και εκεί θέλουμε στενή συνεργασία ώστε να συμμετέχει το Μαρόκο σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα γιατί το θέμα της παιδείας, της μόρφωσης και της κατάρτισης είναι προτεραιότητα και του Μαρόκου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μου απέμεινε πολύς χρόνος, γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω στο τέλος για τη χρηματοπιστωτική συνδρομή και για τις μελλοντικές προοπτικές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική διάσταση της συνεργασίας. Θα ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την συνεργασία σε οικονομικά θέματα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζουμε την επιθυμία η εφαρμογή του προηγουμένου καθεστώτος να ενισχύσει αυτή τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας, αλλά και το δυναμικό απορρόφησης του Βασιλείου του Μαρόκου. Στις συζητήσεις που είχαμε για το Εθνικό Πρόγραμμα 2007-2013 το Μαρόκο επέμεινε στην ανάγκη να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά θέματα και στην ανθρώπινη διάσταση, στο ανθρώπινο δυναμικό. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις επιμένουμε ε, και ζητούμε επίμονα μάλλον την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι σημαντικές οι φιλοδοξίες μας και οι προσδοκίες μας από το προηγμένο καθεστώς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε και νέους πόρους για να συνδράμουμε το Μαρόκο να υλοποιήσει αυτή την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γιατί η βούλησή του είναι δεδουλωμένη, η φιλοδοξία του το ίδιο. Θέλουμε λοιπόν αυτή την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Το επισήμανε προηγουμένω και ο Νέκο Λανταμπούρου Έχουμε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και προσπαθούμε να επινοήσουμε ένα νέο μηχανισμό για να αντικαταστήσουμε το ισχυρό πλαίσιο, ένα μηχανισμό που θα είναι πιο φιλόδοξος και που θα βοηθήσει το Μαρόκο σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη θέσαμε τα θεμέλια μιας πορείας που είναι όλο και πιο φιλόδοξη και μπορεί στο μέλλον να μας οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός νέου μηχανισμού στα πλαίσια αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Τώρα, ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές και οι βασικές προσδοκίες του Μαρόκου. Το Μαρόκο θέλει κυρίως ενίσχυση της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό προσβλέπουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της ε, προχόμενης Ισπανικής Προεδρίας για την έγκριση και τη συγκεκριμενοποίηση μια δέσμη μέτρων. Για παράδειγμα, τη σύσταση μια μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Μαροκινού Κοινοβουλίου, την ενίσχυση και σύσφυξη του διαλόγου, του πολιτικού διαλόγου και σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδων και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης η συνέχιση των εργασιών της ad hoc ομάδας εργασίας για το προηγμένο καθεστώς και η συμμετοχή και νέων φορέων όπως μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, τοπικές αρχές και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά και διάφορα άλλα θέματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα που θα πρέπει να σημειώσουμε πρώτα, όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι ευαίσθητα θέματα, αλλά έχουμε θετική εμπειρία πρόοδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πλέον και τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας και το Μαρόκο είναι πρόθυμο να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει για μια όλο και πιο φιλόδοξη σχέση με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ κύριε και Γραμματεύ. Έχουμε τώρα την παρέμβαση του Διευθυντή Ερευνών του, του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, τον καθηγητή Ιβάν Μαρτίν. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Ε, Θερμά ευχαριστώ σε όλου και κυρίω για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια κρόση, προκειμένου να σα εκθέσω την άποψή μου για το προηγμένο καθεστώ. Ναι και μου το ζητήσετε, θα επικεντρωθώ στα διδάγματα που αντλήσαμε από το προηγμένο καθεστώς με άλλες γειτονικέ χώρες και περιοχές. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τρεις βασικούς άξονες για να αναλύσω αυτή τη διαδικασία διαφοροποίησης που ανέφερε και ο κύριος Σαμπράνη. Θα πρέπει Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε την προστιθέμενη αξία αυτού του προηγμένου καθεστώτος. Τρίτο, να δούμε ποια είναι η συνάφεια αυτού του προηγμένου σχέσεως με άλλα σχέδια προνομιακών σχέσεων με γειτονικέ χώρες και αυτό υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν έρθω όμως στην ουσία του πράγματος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι ένας ανεξάρτητος παρατηρητής και μοναδική μου δέσμευση είναι αυτή η προσήλωσή μου στο στόχο εξασφάλισης ε, χώρου ελευθερίας και ασφάλειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της ε, χωρών. Και ακριβώς επειδή είμαι Ευρωπαίος, θα ήθελα να δώσω έμφαση όχι τόσο στη δέσμευση του Μαρόκου υπέρ του προηγμένου καθεστώτος, ε, που μας παρουσίασαν και ο κ. Ανταμπούλου και ο κ. Αμράνη, αλλά εγώ θα αναφερθώ κυρίως στην ευρωπαϊκή δέσμευση και το τι είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σε θέματα προηγμένου καθεστώτος με τις γειτονικέ της χώρες. Το προηγμένο καθεστώς είναι μια έμπρεκτη εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης, που εμέσως περιλήφθηκε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές χώρες το 2003. Τότε προσδιορίστηκε η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίασης. Και μέσω μιας διαδικασίας συγκριτικών κανόνων και συγκριτικής ανάλυσης ε, ε, λαμβάνεται υπόψη. Σε μια έρευνα που θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες από το Ινστιτούτο για τη Μεσόγειο για την Ευρωμεσογειακή Σχέση και πάνω από 300 εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτής της ε, ένταξης προβαίνουν σε μια πολύ θετική αξιολόγηση αυτή τη έμπρακτη εφαρμογή τη διαφοροποίηση. Το 70% των εμπειρογνωμών θεωρεί ότι είναι σκόπιμη εφαρμογή μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην ευρωμεσογειακή λεκάνη. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια για αυτή, για αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση, γιατί χρειάζονται κάποια κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι τα σχέδια δράσης γυτνίασης. Το μαροκινό σχέδιο έχει 9 προτεραιότητες, 89 στόχους και περίπου 300 δράσει. Είναι αδύνατον από αυτό το σχέδιο δράσης γυτνίασης να καταλήξουμε σε ένα σαφές καλούπι κριτηρίων για να εφαρμόσουμε τη διαφοροποίηση. και άλλα και στα άλλα σχέδια δράσης το ίδιο συμβαίνει. Και όταν εξετάζουμε τις μελέτες πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματικά διευκρινίζουν τις α, σχέσεις γειτνίασης, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι κανονικές εκθέσεις πρόοδου, μια και ουσιαστικά περιγράφουν την κατάσταση, χάρη διαφάνειας, αλλά δεν έχουν ένα στερεότυπο, ένα, ένα συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα. Ούτε έχουν κριτήρια που να επιτρέπουν τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των διαφόρων χωρών ούτε εκπληρώνουν τα ελάχιστα κριτήρια παρακολούθησης ε, και ελέγχου των πολιτικών που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και για πολιτική απασχόληση ή παιδείας που δεν είναι κοινωτικές αρμοδιότητες. Με το Ίδρυμα ΕΒΕΡΤ καταλήγουμε σε 30 ε, προτάσεις για μια μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίηση αυτών των μέσων η πολιτική γετνίασης δεν μας προσφέρει κάποια πρακτικά κριτήρια διαφοροποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε τον Οκτώβριο του 2008 ότι θα πρέπει να γίνει ένα είδος αναβάθμισης των σχέσεων. Αυτό συνέβη με το Ισραήλ. Και λίγες μέρες μετά την δημοσίευση της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ε, έκρινε ότι στα κατεχόμενα εδάφη δεν τηρούνταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρξε πρόταση αναβάθμιση. Δεν υπάρχει σχέση λοιπόν αιτίου και ιδεατού μεταξύ της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της εκθέστης και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτό το ενισχυμένο καθεστώς ή τις προνομιακές σχέσεις ή της αναβάθμισης με το Ισραήλ, που τελικά βέβαια παρεμποδίστηκαν αλλά για άλλους λόγους. Στην περίπτωση του Μαρόκου υπάρχει συνένεση ότι υπήρξε πρόοδος και το προηγμένο καθεστώς αυτό αντικατοπτρίζει αλλά λίγες εβδομάδες μόλις μετά την υπογραφή του κοινού εγγράφου για το προηγμένο καθεστώς, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υποχρεώθηκε να προβεί σε εκτενή δήλωση εξηγώντας τις ε, ε, προνομιακέ σχέσει, ειδικέ σχέσει που θα έχει με άλλε γειτονικέ χώρε όπω ήταν η Τινησία, η Αίγυπτο και η Ορδανία. Ουσιαστικά λοιπόν ε, αλλοιώνει το προνομιακό προηγμένο καθεστώ με το Μαρόκο, γιατί φαίνεται ότι γενικεύει ένα τέτοιο είδο ιδιαίτερη και προνομιακή μεταχείρισης. Δεύτερο στοιχείο τη ανάλυση. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία του προηγμένου καθεστώτος ή πόσο προηγμένο είναι αυτό το προηγμένο καθεστώ, όπω λέει και το άρθρο που σα μοίρασα. Το νέο κριτήριο είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίαση που θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο σχέσεων με όλε τι χώρε, όχι ε, της νότιας, Ευρω... Ε, νότιας της Ευρώπης αλλά και ανατολικά. Ως εκ τούτου, το σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της α, ε, πρόοδου στο προηγμένο καθεστώς είναι αυτό. Και το πιο λογικό θα ήταν το σύνθημα όλα εκτός από συμμετοχή στα θεσμικά όργανα που εξαγγέλθηκε την ίδια ημέρα που υπευλήθη στις Βρυξέλλες το, το προηγμένο καθεστώς. Όταν αναλύσουμε το προηγμένο καθεστώς του Μαρόκου, διαπιστώνουμε ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις σε θέματα πολιτικού διαλόγου. Υπήρξε κάποια πρόοδος και στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή ε, Συνθήκη και Συμφωνία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, αλλά το ίδιο το έγγραφο του προηγμένου καθεστώτος ε, αναφέρεται ως οδικός χάρτης ε, με κάποιες προοπτικές για το Μαρόκο, αλλά χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο. Το μόνο ουσιαστικό περιεχόμενο βρίσκεται στον πολιτικό διάλογο. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τις τρεις Αν ε, πρέπει να δούμε τις τρεις προτεραιότητες του Μαρόκου, ως προσχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλέπουμε ότι είναι η γεωργία, η χρηματοπιστωτική αρρωγή και η διακίνηση των προσώπων. Αυτό φαίνεται από όλε τι μελέτε που έγιναν στο Μαρόκο. Αλλά για αυτού του τρει τομεί δεν υπήρξε καμία πρόοδο. Μάλιστα, το προηγμένο καθεστώ για τη γεωργία να πέμπει στι ε, εκρεμεί διαπραγματεύσει για τη γεωργία. Και στο θέμα τη ε, ελεύθερη κυκλοφορία λέει ότι οποιαδήποτε πρόοδος εξαρτάται ή μάλλον ε, προϋποθέτει την προηγούμενη υπογραφή της Συμφωνίας Επανεισδοχής από το Μαρόκο. Αν το Μαρόκο όμως υπογράψει αυτή τη Συμφωνία, ε, τη συμφωνία Επανεισδοχής, τι αντάλλαγμα θα λάβει. Θα λάβει κάποιο τουλάχιστον καθεστώς διευκόλυνσης ό,τι αφορά τις θεωρήσεις. Δεν αναφέρεται τίποτα. Ή για το θέμα της χρηματοπιστωτικής αρρωγής. Αναφέρεται θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι απαραίτητοι πόροι σύμφωνα με τις φιλοδοξίες του προηγμένου καθεστώτος. Αλλά αναφέρεται ότι μέχρι το 2014 δεν προβλέπεται καμία αλλαγή εξαιτία των δημοσιονομικών προοπτικών. Οπότε να βάλετε η λήψη οποιοδήποτε μέτρου. Από αυτή την άποψη, το προηγμένο καθεστώς σήμερα είναι μία απλή ετικέτα που έχει την αξία του πολιτικού μηνύματος, της δεδηλωμένη βούληση των συμβαλωμένων μερών για πρόοδο, αλλά χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η θέση σε εφαρμογή του προηγμένου καθεστώτος στα πιο ορατά σημεία, όπως είναι η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, θα καθυστερήσει 1,5 χρόνο. Από τις 13 Οκτωβρίου του 2008 που υπογράφει αυτό το κοινό έγγραφο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2010 που θα γίνει η διάσκεψη κορυφής μεσολαβεί 1,5 χρόνος. Κάτι που έρχεται σε αντίφαση με το σχέδιο ε, σύνδεσης Ανατολικής που αμέσως μετά το, την υπογραφή του εγγράφου είχαμε μέσα σε λίγες εβδομάδες τη διάσκεψη κορυφής, ενώ στην περίπτωση του Μαρόκου υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Το Συμβούλιο στην ανακοίνωση του 2008 αναφέρεται κάτι για τις ειδικέ προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ ή με την Ιορδανία και την Ισία. Και η Ανατολική Συμφωνία Σύνδεσης είναι παρόμοια με αυτό το προηγουμένο καθεστώτος. Βέβαια, η, η Ανατολική Συμφωνία Σύνδεσης είναι πολυμερής, ενώ το προηγμένο καθεστώς είναι διμερές. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλε διαφορέ δεν υπάρχουν. Αναφέρεται η ευρωπαϊκή πολιτική γυτνίαση που συνοδεύεται από έναν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. Και μάλιστα δίνεται πολύ μεγαλύτερη σημασία στον πολιτικό διάλογο γίνεται εμβάθυνση και διεύρυνση των ε, ζωνών ελευθέρου εμπορίου, εμπορίου που περιλαμβάνουν και εμπόριο, γεωργία κτλ. και υπογράφεται μια νέα συνθήκη ή μια νέα συμφωνία με τις γειτονικές χώρες. Και όλα αυτά ε, επανέρχονται σε όλες τις ε, συμφωνίες ενισχυμένων σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές της χώρες και όχι μόνο στο προηγμένο καθεστώς. Οπότε έρχομαι στο τρίτο στοιχείο της συζήτησης που είναι η συνάφεια και η συνοχή όλων αυτών των πρωτοβουλειών. Για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή, που δεν συμμετείχε δηλαδή στη χάραξη αυτών των πολιτικών, δεν φαίνεται αυτή η συνοχή, η συνάφεια. Δεν λέω ότι είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχουν πολιτικά έγγραφα που να προβλέπουν αυτή τη συνοχή, τη συνάφεια και η συνάφεια μεταξύ στόχων και μέσων ή μέσω των διαφόρων ε, ε, προνομιακών σχέσεων με το προηγμένο με το προηγμένο καθεστώ για το Μαρόκο, με την Ανατολική Σύνδεση, με τις προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ και τη διαπραγμάτευση με την Τινησία, δημιουργείται μία σύγχυση μεταξύ όλων αυτών των ε, μέσων συνεργασίας. Μία σύγχυση και μία έμεση διάκριση μεταξύ της Ανατολικής Σύνδεσης και της χώρες νοτίου της Μεσογείου. Στην περίπτωση της Ανατολικής Σύνδεσης είχαμε κινητοποίηση 650 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είναι πολλά βέβαια για 6 χώρες, αλλά στο Μαρόκο δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ. Επίσης, τέσσερις θεματικές πλατφόρμες που ε, κινητοποιήθηκαν για την Ανατολική Σύνδεση δεν έχουν καμία αντιστοιχεία με την πρόταση προηγμένου καθεστώτος για το Μαρόκο. Το θέμα της διευκόλυνσης των θεωρήσεων η διευκόλυνση στην πρόσβαση αγοράς εργασίας που αναφέρεται στην Ανατολική Συμφωνία Σύνδεσης δεν αντιστοιχεί σε τίποτε παρόμοιο στο προηγμένο καθεστώς για το Μαρόκο. Ούτε στην ενίσχυση των θεσμικών οργάνων υπάρχει τέτοια αναφορά στο προηγμένο καθεστώς. Είναι πολύ πιο έντονα όλα αυτά τα σημεία στο θέμα της, ε, στη Συμφωνία ε, Ανατολικής Σύνδεσης από ότι στη Συμφωνία με το Μαρόκο. Πώς θα βάλουμε μία τάξη σε όλες αυτές τις συμφωνίες ε, που είναι πολύ συγκεχημένες και ακατανόητες για τον απλό πολίτη. Είναι δυσνόητες ακόμη και τους εμπειρογνώμονες όλες αυτές οι συμφωνίες, αυτή η πληθώρα των συμφωνιών που δίνουν σάρκα και οστά στην πολιτική γειτονία. Περιμένουμε βέβαια την πρώτη διάσκεψη κορυφής με το Μαρόκο που θα γίνει το Μάρτιο του 2010. Φαντάζομαι θα δοθεί πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στο προηγμένο καθεστώς με τη διάσκεψη αυτή κορυφής και μια πιο συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία. Και χρειαζόμαστε και μια γενικότερη εστίαση, ώστε να συνδυαστούν οι εξελίξεις σε συγκεκριμένους τομείς με ενάυσματα σε αυτούς τους τομείς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχέση του μεταξύ προόδων, κανονιστικών ρυθμίσεων και εναυσμάτων σε συγκεκριμένο τομέα. Γίνεται μια γενική αξιολόγηση όλων των κλάδων που αφορά η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αλλά δεν υπάρχει σύνδεση ε, μεταξύ της αξιολόγησης και των εναυσμάτων και των κινήτρων. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες δέσμες ε, παραχωρήσεων που να ισχύουν για όλες τις χώρες της πολιτικής γειτονία. Και θα επιτρέπουμε μια διαφοροποίηση των σχέσεων που θα ξεκινάει από μια συμφωνία σύνδεση όπως αυτή που θα υπογράψει η Αλγερία που θα είναι η ελάχιστη συμφωνία ή με τη Λιβύη κάτι ακόμη πιο ίσονα σημασία, έω τον πραγματικό στόχο που είναι όλα εκτό από τα θεσμικά όργανα. Και από σημειολογική άποψη, όλα εκτό από τα θεσμικά όργανα σημαίνει συμμετοχή και στην κοινή γεωργική πολιτική, συμμετοχή και στην περιφερειακή πολιτική, που είναι οι πιο σημαντικέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ, γιατί αυτό σημαίνει όλα εκτό από του θεσμού. Και αυτό υποσχέθηκε στο Μαρόκο το, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, προβλέπεται και ένα ε, πλέγμα σχέσεων μεταβλητής ε, γεωμετρίας. Χώρες όπως την Ισία που δεν μπορούν να έχουν ε, ευρυθεί συνεργασία ή δεν είναι δεσμευμένα για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι δεν θα ευαθηθούν οι σχέσεις στους τομείς που είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Πάντως είναι επίγον να βάλουμε μια τάξη σε όλο αυτό το πλέγμα των συμφωνιών που αυτή τη στιγμή για τους περισσότερους συμπειρογνώμενους και για μένα δεν είναι της αρεσκίας μας. Σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, έχω σημειώσει κάποιους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Θέλω να χαιρετήσω και να πω ότι είναι παρούσα μια αντιπροσωπεία του Ευρωμεσογειακού Δικτύου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρτίζεται από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων του Μαρόκου και στην είσοδο είναι διαθέσιμη μια έκθεση που συντάχθηκε από αυτό το δίκτυο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της γειτονίας, ε, σχέσεων γειτονίας Ευρωπαϊκής Ενώσης με Μαρόκο. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Άτκινς και του δίνω το λόγο. Πρόεδρε, Είμαι ο μόνος που ήταν εδώ από την αρχή και γι' αυτό έχω μία-δύο σύντομες ερωτήσεις. Πολλοί με... Τρία λεφτά είπατε. Α, <laughs> πολλοί με ικανοποίησαν οι εισηγήσει που έγιναν από τους τρεις ομιλητές με τις διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν και πραγματικά είναι διάφορες οι απόψεις. Θα ήθελα να ρωτήσω Εάν, ποιο είναι το όφελος όλης αυτής της ιστορίας. Κάποιο όφελος δεν υπάρχει, κάποιο κέρδος, αν είναι πολιτικό ή οικονομικό ή κοινωνικό. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν οι τρεις προλαλήσαντες Ομιλούν εδώ περί μιας ε, διοικητικής ε, συμφωνίας, διοικητικής ρύθμισης ή εάν υπάρχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πω για το Μαρόκο όσον αφορά τις πολιτικές επιπτώσεις. Το Μαρόκο προσπαθεί να εδραιώσει σχέσεις στο σημείο, δηλαδή στο παραπέντε πριν από το σημείο ένταξης. Σχέσεις οι οποίες να είναι ε, πλήρεις αλλά όχι ενταξιακές. Παραδείγματο χάρη όμως, τι γίνεται τώρα με την περίπτωση την αμφιλεγόμενη της Τουρκίας, αν γίνει όχι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως λοιπόν ένα παρόμοιο τέτοιο πλαίσιο σχέσεων μπορεί να γίνει και με την Τουρκία. Και το πρόβλημα της ε, παράνομης της μετανάστευσης. Έχει συζητηθεί το μεταναστευτικό και εάν όχι θα συζητηθεί και τέταρτον, ε, ποιες είναι οι οικονομικές σχέσεις του Μαρόκου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι επιπτώσεις υπάρχουν σε, αυτό, σε αυτές τις οικονομικές ρυθμίσεις. Και πέμπτον και τελευταία ερώτηση, αποτελεί αυτό προηγούμενο αυτή η ρύθμιση και για άλλες ε, περιπτώσεις εν συνεχεία με άλλες χώρες ή είναι μια εξαιρετική περίπτωση αυτή η ρύθμιση με το Μαρόκο που δεν θα επανελειφθεί για άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Η κυρία Στράσερ, παρακαλώ. Ο κύριος Στράσερ, συγγνώμη, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να συγχαρώ ακόμα όλους αυτούς ε, που βοηθούν ε, σε μια τέτοια προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως αυτή η προσπάθεια, διότι οι μεσογειακές χώρες έχουν ιδιάζουσα σημασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι αυτών των χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμπεριλάβει γειτονικέ χώρες ε, της Μεσογείου με, μια πολύ ε, συνετή μορφή, με ένα πολύ καλό τρόπο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε προς το παρόν όλους αυτούς που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έχω μια ερώτηση η οποία συνάδει με την Συμφωνία για την Ασφάλεια και την Επαναφορά το, το δίκτυο επαναφορά, το ρεφουλμό, ε, τι θα γίνει με αυτή την ε, περίπτωση και αν έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ τον κύριο Στράσε ή συνάδελφος ο Ιουλάντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να... Ε, συγχαρώ τους προ... όλους όσους συνέδραμαν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στους συναδέλφους από το Μαρόκο. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα ε, για τις... Ε, τα βήματα πρόοδου που έχετε επιτύχει μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, πιστεύω ότι έχετε προσεγγίσει την, την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε σύντομα να συμμετάσχετε και σε άλλους φορείς. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Λανταμπούρου. Υπάρχουν προοπτικές ε, μεταξύ Μαρόκου και Ένωσης ε, ενίσχυσης ε, της ενεργειακής συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας για την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Κύριο... Το λόγο δίνω στο συνάδελφο Μπεν Αραμπ, στο συνάδελφο στη συνάδελφο Μπελαράβ. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Αμράνη έχω ένα ερώτημα. Πώς θα διαρθρώσετε τη συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή, με, τις, με τους συνεργάτες σας του Μαγκρέμπ, του Αραβικού. Μια πραγματική ένταξη στο Μαγκρέμπ που, που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Μια ένταξη πραγματική ενοποίηση στο πλαίσιο του Μαγκρέπ θα επιτρέψει πιο ισορροπημένη διαπραγμάτευση στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Η τελική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως με μια πραγματική ένωση του Μαγκρέπ δεν είναι καλύτερη παρά να γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως με κάθε χώρα του Μαγκρέπ. Κατακαιρματισμένα και λιγότερο ισορροπημένα. Ταυτόχρονα θέλω να αναφορθώ στο μεγάλο συγγραφέα, τον Αμπτέλ Κιμπίρ Χατιμπή και το έργο του το ε, Μαγκρέπτο. δεύτερο ερώτημα αφορά όλους όσους πήραν το λόγο. Προτίθεστε να βρείτε μια λύση για τη διαθέτηση του δρόματος των ε, νέων μεταναστών από τη νότια, τις νότιες ακτές Μεσογείου που πολύ συχνά προσπαθούν να πάνε στις βόρειες ακτές και πνίγονται συχνά. Χρειάζεται συνεργασία, γιατί σωρεύονται τα πτώματα στη Μεσόγειο λόγω αυτού του προβλήματος. Χρειάζεται γρήγορη λύση. Ποια μπορείτε να φανταστείτε που μπορείτε να εφαρμόσετε λύση, πραγματική κινητικότητα δεν θα δημιουργείς πιο ανθρώπινες προπτικές για όλους αυτούς τους ε, νέους. Ευχαριστώ, κυρία Μπεναράμπ. Για να δώσουμε ώρα σε όλους, σας παρακαλώ να είστε συνοπτικοί στις παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Αγκουράκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σημειώσω ότι η ομάδα Γκουε όταν έγινε συζήτηση για αυτή την πρωτοβουλία είχε ζητήσει να υπάρχει και εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σαχράουη. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι σήμερα δεν βρίσκεται κανείς εκπρόσωπός τους μαζί μας. Δεύτερον, θα ήθελα να σημειώσω ότι εγώ, εμείς τασόμαστε ενάντια στο Advanced Status ε, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο και αυτό γιατί κατά τη γνώμη μας υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά αφορά τόσο το εσωτερικό της χώρας όσο και τα εξωτερικά ζητήματα, κυρίως το ζήτημα ε, της ε, Δυτικής Σαχάρας όπου ε, το Μαρόκο ε, καταπατεί το διεθνές δίκαιο και δεν εφαρμόζει αποφάσεις του ΟΗΕ. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής τον κύριο εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πρώτον, τι σκέφτεται να κάνει η Κομισιόν ώστε το Μαρόκο να σεβαστεί επιτέλους τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σταματήσει την καταπίεση ενάντια σε υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Δεύτερον, ποια είναι η θέση της Κομισιόν σχετικά με την αντιπαράθεση και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας και τρίτον και τελειώνω με αυτό ε, αναρωτιέμαι εάν η Κομισιόν γνωρίζει την υπόθεση της κυρίας Χαμινάτου Χαϊντάρ, αγωνίστρια Σαχραουή. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνει η Κομισιόν ώστε το Μαρόκο να επιστρέψει στην κυρία Χαϊντάρ το διαβατήριό της και να της δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη χώρα της. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Κύριος Ρομέρο Λόπες έχει το λόγο. Η κυρία Ρομέρο Λόπες. Eh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Αμράνη, τον πρέσβη Λανταμπούρ, τον κύριο Μαρτίν. Χαίρομαι που ήρθατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που για μας τους Ισπανούς είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανάλυση που μας κάνατε της προστιθέμενης αξίας αυτού του προηγμένου καθεστώτος. Αυτό είναι σημαντικό για να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως υπόδειγμα για συμφωνίες σύνδεσης με άλλες χώρες. Αναφέρθηκε η Ανατολική Συμφωνία σύνδεση. Και είχαμε μια εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας προς Ανατολάς. Και έχουμε προς Ανατολάς κάποιες προτεραιότητες, αλλά πέραν τούτου το προηγμένο καθεστώς προϋποθέτει την δημιουργία ενός ιστού διασυνδέσεων που είναι πολύ σημαντικές, ώστε να μην έχουμε μια αμυγή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή αμυγή εμπορική συμφωνία. Θέλουμε μια πολυδιάστατη συμφωνία που δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά και πολιτική, κοινωνική, ανθρώπινη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα στο σχέδιο δράσης του κοινού εγγράφου αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα και προβλέπεται διάλογος με μη κυβερνητικέ οργανώσεις ώστε από αυτό τον κοινό διάλογο με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο βήμα, αλλά εκρεμεί και η συμφωνία σύνδεση με τη Λιβύη. Και εκεί μένει να δούμε τι μοντέλο θα διαλέξουμε, αν υιοθετήσουμε ένα παρόμοιο μοντέλο με αυτό που έχουμε. Και δεν λέω για την Ιορδανία και την Τινησία. Καλό θα ήταν και στις συμφωνίες αυτές να ασχοληθούμε με τους τομείς που καλύπτει και το προηγμένο καθεστώς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κατεύθυνση και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο βήμα μόνο. Θα πρέπει όμως στη συνέχεια να γίνει αξιολόγηση. Κύριε Λανταμπούρου, θα γίνει κάποια αξιολόγηση αυτού του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προηγμένου καθεστώτος. Έγινε μια τέτοια αξιολόγηση του πρώτου χρόνου εφαρμογής. Εντοπίστηκαν κάποιες δυσκολίες που δεν αναφέρθηκαν στις ομιλία σας, για παράδειγμα, στις υπηρεσίες ή σε έναν άλλο τομέα. Και εκεί ίσως θα μπορούσαμε εμείς οι ευρωβουλευτές να συμβάλλουμε για την ε, ομαλή διεξαγωγή κάποιων σημείων του καθεστώτος. Στο Κιλ Νίλσεν είναι το επόμενο όνομα που έχω στον κατάλογο. Κυρία Κιλ Νίλσεν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω επί ενός θέματος που εφήγη προηγουμένως και γι' αυτό ζήτησα να πάρω το λόγο μια συζήτηση για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Μαρόκου, πιστεύω ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα σοβαρά χωρί να θέσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίω το θέμα τη Δυτική Σαχάρα. Οι κάτοικοι τη Σαχάρα υπόκεινται σε, μια, σε καθημερινό επικισμό και ταπεινώσει. Προ... Συλλαμβάνονται οι ειρηνικοί αντιπολιτευόμενοι, πολλαπλασιάζονται συλλήψει του τελευταίου μήνε. Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει η Ευρώπη, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να εγγυηθεί το δικαίωμα των κατοίκων της Σαχάρας για αυτοδιάθεση, σεβόμενοι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και θα ήθελα, όπως και κάποια συνάδελφος προηγουμένως, να αναφερθώ στο θέμα ε, για στην αμήνα του ΑΙΔΑ που απελάθη στις 14 Νοεμβρίου από τη χώρα της που είναι σε απεργία πείνας εδώ και τις εβδομάδες και είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μη Μηπω θα πρέπει να το θέσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συζητήσει και κυρίως στην ε, Δυτική Σαχάρα πιο συγκεκριμένα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νίλσεν. Επόμενο όνομα, Σόλτ. Ο κύριος Σόλτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ είχα ζητήσει το λόγο γιατί με ενδιαφέρουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί, αλλά τώρα έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα απευθύνουμε στην Κομισιόν και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε την προοδευτική αυτή συμφωνία τμήμα της Μεσογειακής Ένωσης και της Μεσογειακής Πολιτικής. Και τι προτεραιότητα δίνει σε τέτοιου είδες συμφωνίες. Το δεύτερό μου ερώτημα είναι πώς θα χειριστεί τις προβληματικές σχέσεις μεταξύ μεσογειακών χωρών όπως το άλυτο πρόβλημα του Μαρόκου και της Δυτικής Σαχάρας. Πιστεύω ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στη λύση αυτού του προβλήματος στο άμεσο μέλλον για να βοηθήσουμε σε μια καλύτερη εδραίωση μιας ολοκληρωμένης μεσογειακής πολιτικής. Μήπως θα μπορούσατε και οι εκπρόσωποι του όσοι μίλησαν από πλευράς Μαρόκου να απαντήσουν. Σας ευχαριστώ. Φλέτχο, επόμενο όνομα που έχω. Κυρία Φλέτχο, κλείνει τον κύκλο. Αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στο προωθημένο, στο ενισχυμένο καθεστώ των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου. Αυτό θεωρείται ότι η χώρα αυτή είναι σε προνομιούχα θέση, αλλά βέβαια τίθεται και διάφορα ερωτηματικά εφόσον αυτή η πρώτη χώρα, που αφορούν λιγότερο την κατάσταση που κρατεί στο Μαρόκο παρά τη μεθοδολογία και του μηχανισμού που θέλει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να νομιμοποιήσει, να δώσει ουσία στο ενισχυμένο αυτό καθεστώ. Είδαμε τη συζήτηση στα πλαίσια τη επαναπρόθεση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ενώσεω Ισραήλ που πάγωσαν σχέσει κατά τη διάρκεια των σειράξεων στη Γάζα και το Συμβούλιο βρήκε υπεκφυγή να μην δώσει σύμφωνη γνώμη στο θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ στις διάφορες κοινοτικές υπηρεσίες. Ερώτημα για να βρούμε κάτι που να οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα στα πλαίσια του ενισχυμένου καθεστώτος. Πολλοί αναφέρθηκαν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημοκρατία. Σημαντικό θέμα. Αλλά θέμα αξιολόγησης και συμμετοχής των πολιτών τίθεται μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων και βουλευτών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτω το ερώτημα. Πώς να το πω, υπάρχουν εκ των προτέρων κριτήρια που θα μπορούσαν να μοιάζουν με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Ένα είδος κριτήρια Κοπενχάγης για να ξεκινήσει η εφαρμογή του νησημένου καθεστώτος. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Αύριο θα δώσουμε το καθεστώς αυτό στην Τινησία, παραδείγματος χάρη, που φυλακίζει κόσμο και απειλεί τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παίξουν ρόλο. Υπάρχουν πολύ σημαντικά μεταίσθηση δικαστικού τομέα κατά στις φυλακές τι γίνεται, η δίωξη διαφόρων φορέων προστατεύοντα τα δικαιώματα, καθεστώ των προσφύγων. Αυτά τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση για το Μαρόκο, πόσο βάρο έχουν, πόσο μετράνε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πότε θα πρέπει να πούμε κάτι, πέρα από αυτού του είδου ακράσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ποια κριτήρια εφαρμόζονται Ποιο οδικό χάρτη θα ακολουθηθεί, ποιο μηχανισμό που θα μα επιτρέψει να εφαρμόσουμε πραγματικά και να ελέγξουμε την εφαρμογή του δικού χάρτη από την έποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία. Το θέτω για το Μαρόκο μεν, αλλά εγώ θέλω να έχουμε ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιόπιστους και διαφανείς που θα μα επιτρέπουν πραγματικά ω ευρωβουλευτέ να παρεμβαίνουμε όσον αφορά την εφαρμογή, το περιεχόμενο, το πότε ξεκινάνε να ενισχύουν τα καθεστώτα, πώ εφαρμόζονται και αξιολόγηση του καθεστώτος αυτού. Διαφορετικά δεν ξέρω τι ακριβώ ακολουθεί μετά την εφαρμογή του ενισχυμένου καθεστώτος. Ευχαριστώ κυρία Φλότρο. Θα δώσω το λόγο στους εισηγητέ, παρακαλώντα του ή δυνατόν να παραμείνουν στο πεντάλεπτο. Και θα ακολουθήσω αντίστροφη σειρά. Να δώσω πρώτα το λόγο στον καθηγητή Μαρτίν και μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Αμράνη και μετά ο επικεφαλής αντιπροσωπείας κ. Λανταμπούρου. Επιγραμματικά έξι παρατηρήσεις για τη μετανάστευση που ανέφερε κάποιος Άγγλος Ευρωβουλευτής και κάποιος Γερμανός. Δεν γνωρίζω τα ονόματά τους. Συμφωνία επανεισδοχής. Το Μαρόκο φαίνεται δεν είναι δετεθειμένο να υπογράψει αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής που είναι σημαντική για την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καλή αυτή η διαπραγματευτική στρατηγική να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψτε εσεί τη Συμφωνία Επανεισδοχή και μετά θα αρχίσουμε τι διαπραγματεύσει. Κάποιο αντάλλαγμα θα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, με τι χώρε τη Νοτιού Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ούτε καν να δώσει προοπτική διευκόλυνση του καθεστώτο θεωρήσεων. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και από την άποψη ε, κινητικότητα, ελεύθερη διακίνηση, ε, συνιστά διακριτική μεταχείριση ανατολικών χωρών και νότιων χωρών. Ούτε θα πρέπει να ζητούμε Ω απαραίτητη προϋπόθεση τη Συμφωνία πανιστοχή. Δεύτερον, το προηγμένο καθεστώ έχει και πολιτικέ ε, επιπτώσει. Δεν είναι μία απλή διοικητική εφεύρεση. Οι πολιτικέ επιπτώσει βέβαια θα είναι πιο χρονοβόρε στην εφαρμογή. Αλλά εδώ μιλούμε για την αρχιτεκτονική των σχέσεων με τι άλλε χώρε που δεν θα είναι γειτονικέ. Και από αυτή την άποψη η έκφραση όλα εκτό από του θεσμού προήλθαν από τι διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά αυτός ο όρος από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Ρωμάνο Πρόντι. Αν δεν υπάρχει, αν δεν γινόταν ένταξη της Τουρκίας, το όλαχο εκτός από τους θεσμούς θα ήταν ε, η εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος σύγκλησης μεταξύ των σχέσεων που υιοθετήσαμε με την Τουρκία και των προνομιακών σχέσεων με τις άλλες χώρες. Τρίτον, το προηγμένο, το ενισχυμένο αυτό καθεστώς παρόλο που αναφέρεται ως κάτι συγκεκριμένο για το Μαρόκο, δεν ισχύει. Υπάρχει ένα είδος καλουπιού, υπάρχει ένα κοινό καλούπι, εκμαγείο μεταξύ του, του προηγμένου καθεστώτος, του ενισχυμένου καθεστώτος, της ανατολικής σύνδεσης και της πρώτης αναβάθμισης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και από αυτή την άποψη φαίνεται ότι βαδίζουμε προς ένα νέο μοντέλο σύσφυξης σχέσεων. Και είναι ενισχυτικό το γεγονό ότι γίνεται χωρί ε, ε, συγκεκριμένη πολιτική διαδικασία και χωρί ένα ιδρυτικό έγγραφο που θα προσδιορίζει του στόχου, τα μέσα κτλ. Τέταρτο, πέμπτο θέμα. Η Ένωση Αραβικού Μαγκρέμπ. Δεν ήταν για μένα η ερώτηση, αλλά το θέμα αυτό είναι κέριο. Όχι μόνο για την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, αλλά για την ε, συνεργασία στο Νότο. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν ε, της διένεξης της Σαχάρα, που όντως ε, μπλοκάρει τις σχέσεις ε, Αλγερίας-Μαρόκου, αλλά δεν είναι η αιτία του αδιεξόδου. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις, τη συνεργασία του Νότου μεταξύ των χωρών του Μαγκρέπ. Με την Αλγερία μιλούν κυρίως για ενέργεια, για ελεύθερη διακίνηση, αλλά τίποτα δεν αναφέρεται για την ένταξη και την ολοκλήρωση στις χώρες του Μαγκρέμπ. Δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα. Δεν λέω ότι θα πεμπλέξει τα πράγματα, αλλά ούτε αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Το θέμα της κοινωνίας των πολιτών που επισήμανε η κυρία Ρομέρο είναι πολύ σημαντικό. Και από αυτή την άποψη το κοινό έγγραφο του ενισχυμένου καθεστώτος θα μπορούσε να είναι χρήσιμο έγγραφο και χρήσιμο μηχανισμός προώθησης των σχέσεων μεταξύ των ε, τοπικών αυτοδιοικήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, για να δημιουργηθεί αυτός ο ιστός και η διασύνδεση που είπατε. Επίσης, ε, ήδη εφαρμόστηκαν κάποια στοιχεία του ενισχυμένου καθεστώτος, όπως η συμμετοχή σε συγκεκριμένες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Από ό,τι ξέρω δεν έγινε τίποτα συγκεκριμένο στα πλαίσια του ενισχυμένου καθεστώτος για να ε, συσφιχθούν οι σχέσεις μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ήδη υπήρχαν κάποιες σχέσεις, αλλά δεν αναπτύχθηκαν. Ούτε μεταξύ των τοπικών ή περιφερειακών αυτοδιοίκησεων ενισχύθηκαν οι σχέσεις. Οπότε από αυτή την άποψη τη προστιθέμενη αξία μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Με το Μαρόκο υπογράφηκε το ενισχυμένο καθεστώς, ο δικός χάρτης δηλαδή. Με το Ισραήλ όμως μην ξεχνάτε ότι στις 15 Απριλίου του 2008 υπογράφηκε πρωτόκολλο με συμφωνία πλαίσιο για συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής για το Μαρόκο, οπότε είναι σαφές ότι δεν είναι το Μαρόκο η πρώτη χώρα με την οποία ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προνομιακή σχέση. Με το Ισραήλ είχε ακόμη πιο προνομιακή. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε τις, φήμε φήμες ότι έχουν αρχίσει συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις με την Τινησία με απότερο σκοπό να συμφωνηθεί ένα, ενισχυμένο καθεστώς σχετικά σύντομα. Θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός για να αποσυνδεθούν οι πρόοδοι στους διάφορους, ε, σε στο σύνολο των τομέων ώστε να προωθηθεί η εξέλιξη σε ορισμένους τομείς. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προηγουμένο ενισχυμένο καθεστώ στην Τινησία χωρί προηγουμένω να διευκρινίσει τα κριτήρια τη Κοπεχάγη, των Βρυξελών για τη σχέση με τι τρίτε χώρε που μέχρι στιγμή αυτά τα κριτήρια είναι ασαφή και συγκεχημένα. Σα ευχαριστώ. Υπήρξατε πλήρη και σύντομο στην παρέμβασή σα. Ο Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών έχει το λόγο τώρα. Ο κύριο Αμράνη. Πολλές ερωτήσεις μου τέθηκαν. Θα αρχίσω καταρχάς με την ε, συμφωνία αυτή και αν αποτελεί σημείο προόδου των σχέσεων ε, Βορρά-Νότου. Ναι, βεβαίως αποτελεί ένα βήμα πρόοδου, δεδομένου ότι το Μαρόκο είναι μια χώρα του Νότου. Μας ε, ενδιαφέρει η δική σας εξέλιξη, μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι νέες αγορές, μας ενδιαφέρουν καινούργιες προσπάθειες. Είναι μια φιλοδοξία αυτή του Μαρόκου. Μια φιλοδοξία την οποία έχουμε εκφράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εάν σήμερα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο προηγμένο, αυτό δείχνει ότι έχουμε επιτύχει πολλά όσον αφορά τις κοινέ αξίες, τον διάλογο, την επιτυχία του διαλόγου και την καλή εμπειρία που έχουμε με, με τις σχέσεις μαζί σας στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς. Σήμερα μπορώ να πω ότι το Μαρόκο γνωρίζει εις βάθος τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι ήταν μια αμοιβαία φιλοδοξία αυτή μεταξύ των δύο μερών του Βορρά και του Νότου, της Ευρώπης και ημών. Η Ευρώπη όχι μόνο ενδιαφέρεται, αλλά θέλει και ενεργά να ενισχύσει τις σχέσεις της περαιτέρω με τους νότιους μεσογειακούς γείτονες. Ε, σήμερα το Μαρόκο ε, και το Μαγκρέμπ γενικότερα, σε ευρύτερο πεδίο δηλαδή, αποτελεί μια προτεραιότητα για την Ευρώπη. Όχι μόνο στο πλαίσιο της ασφάλειας, αλλά και στο πλαίσιο της ειρήνης και της σταθερότητας. Διότι ο μεσογειακός χώρος, η Βόρεια Αφρική, είναι γειτονική σας περιφέρεια και για λόγους ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν ειρηνικά δημοκρατικά καθεστώτα και γι' αυτό ακριβώς το Μαρόκο εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και θέλει να ενισχύσει σε κάθε πτυχή την συνεργασία με την, οικονομική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω τώρα με την οικονομική χρήση και στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης χρειάζονται περισσότερες ε, αγορές. Και το Μαρόκο ε, ε, έχει προχωρήσει ενεργά σε όλους τους οικονομικούς τομείς και στον χρηματοπιστωτικό, διότι παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες και δίκερδοφόρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ρωτήσατε, η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει ένα προηγούμενο, ένα μοντέλο. Εμείς δεν θέλουμε να ενεργήσουμε ως μοντέλο, ε, αλλά εάν αυτό το πείραμα επιτύχει μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα στις άλλες γειτονικέ χώρες του Νότου. Σε κάθε περίπτωση το Μαρόκο κάνει τις δικές του μεταρρυθμίσεις. Θα μιλήσω αργότερα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ε, να πορευόμαστε στον δρόμο της δημοκρατίας, στο, δρόμο ε, της ε, ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτός ο δρόμος και επιστροφή δεν υπάρχει. Θα προχωρήσουμε μπροστά και γι' αυτό έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια σε να εδραιώσουμε βασιές πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Σήμερα Σημερίζουμε μαζί σας με αυτό το σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημερίζουμε αυτή την εμπειρία. Δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ, δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό να συζητήσουμε μαζί σας σε βάθος αυτές τις λίγες ευαίσθητες ε, πτυχές, τα πολύ ευαίσθητα θέματα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της μετανάστευσης, ναι, είναι δύσκολο, έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, όποιος ο Μαροκινός βρίσκεται παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος, ε, επανεισέρχεται, ε, υφίσταται τη διαδικασία επανεισδοχής. Το πρόβλημα είναι με τη Δυτική Σαχάρα. Έχουμε κάνει πολλαπλές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή και ποτέ δεν έχουμε ε, συζητήσει αυτό το θέμα και ολοκληρώσουμε το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία η οποία όμως να μπορεί να εφαρμοστεί ε, να είναι δηλαδή ε, λειτουργήσιμη και πολιτικά αποδοκτή. Έχουμε την κοινωνία των πολιτών στην, στο Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν είναι μόνο μια χώρα τράνζιτ όπου διέρχονται ε, άνθρωποι, αλλά έχουμε, βρισκόμαστε και στα σύνορα, αν θέλετε, της Ευρώπης και είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε προς, ποιος προέρχεται από εκεί ή όχι. Το Μαρόκο δεν μπορεί από μόνο του να λύσει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούμε μόνοι, μόνοι μας να φορτωθούμε το τεράστιο βάρος της υποσαχάριας μετανάστευσης. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα καθορισμού του ποιος προέρχεται από ποια περιοχή υποσαχάρη και ποιος όχι. Πράγματι το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και το να πιάσουμε και να σταματήσουμε αυτά τα δίκτυα της ε, παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου ανθρώπων είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν μπορούμε από μόνοι μας να το λύσουμε έχουμε αναγνωρίσει και, γνωρί... και, και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα υπάρχουν στην απόδειξη στο βάρος της απόδειξης. Ποιος μπορεί να αποδείξει ότι αυτό το άτομο προέρχεται όντως από το Μαλή ή τη Σενεγάλη και είναι παράνομα διερχόμενος ή παράνομος με, με, την μετανάστευση. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε το 13ο γύρο διαπραγμάτευσης. Πράγματι είναι προτεραιότητα για το Μαρόκο η ολοκλήρωση στα πλαίσια του Μαγκρέμπ. Πρώτα απ' όλα διότι και ο λαός το θέλει αυτό. Μετά το η ένωση του Μαγκρέμπ είναι στρατηγική αναγκαιότητα για την μετώπιση των διαφόρων επιταγών ασφαλείας, αναπτύξεως κλπ. Και μετά είναι και μια δυνατότητα που δεν πρέπει να χάσουμε, μια ευκαιρία. Δεν θα καταλογίσω ευθύνε σε συγκεκριμένε χώρε όσον αφορά την έλλειψη προόδου για την ε, ολοκλήρωση στα πλαίσια του Μαγκρέμπ αλλά καταδικάζω ότι είναι κλεισμένα κάποια μεθοριακά σημεία που δεν υπάρχει βούληση προφανής των γειτόνων μας να δημιουργηθεί το Μαγκρέπ για λόγους που γνωρίζετε. Ήρθα σήμερα για να μιλήσω για το ενισχυμένο αυτό καθεστώς. Αλλά πώς μου δίνετε ευκαιρία το Μαγκρέπ, από δύο λόγια. Το Μαγκρέπ είναι μια μεγάλη αναγκαιότητα, επιτακτική ανάγκη, θα πρέπει να γίνει το Μαγκρέπ, διότι ακόμα και για την Ευρώπη είναι ενδιαφέρον, συμφέρον, υπάρχει ε, ένας φορέας που να μπορεί να συνομιλεί με την Ευρώπη συγκεκριμένα θέματα ασφαλείας, οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βασιστείτε στο Μαρόκο, δεν θα αφιστεί προσπαθειών, ούτω ώστε να, βάλει, να θέσει ξανά στην τροχιά τη σωστή το πρόγραμμα για το Μαγκρέμπ. Είναι προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Το Μαρόκο όχι μόνο είναι αποφασισμένο, αλλά μεριμνεί ούτως ώστε αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεω με το Μαγκρέπ να αποκτήσει χτίσει μια υφή. Και στο Ραμπάτ ε, οργανώθηκε η πρώτη συνεδρίαση μεταξύ Τρόικα Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των χωρών του Μαγκρέπ του Αραβικού για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίε για την δημιουργία του Μαγκρέπ. Παραμένουν οι δυσκολίε, χρειάζεται δουλειά για να δημιουργηθεί το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών του Μαγκρέπ. Το Μαρόκο είναι αποφασισμένο να κάνει το καθήκον του σχετικά με αυτό το θέμα. Α, αμέσως, αμέσως, ναι. Θα μιλήσω ισπανικά τώρα. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήθελα να το θίξω εγώ σήμερα. Γιατί άλλο το αντικείμενο της σημερινής ακρόασης είναι το, προ... το ενισχυμένο καθεστώς. Αλλά με καλέστε να μιλήσω για ένα θέμα που είναι πολύ ευαίσθητο. απόψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδημοκρατισμού, το Μαρόκο δεν έχει κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας. Είμαστε η μοναδική χώρα της περιοχής που έχει Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνέρχεται τακτικά για να εξετάσει όλα τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα όμως της Σαχάρας της Μαροκινής δεν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν υπάρχει εδώ θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μαροκινική Σαχάρα. Και μάλιστα ειδικό επισταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εντατικοποιεί τι προσπάθειε του προκειμένου να διεκπαιρεθεί και δεύτερη άτυπη συνεδρίαση με στόχο την ενίσχυση των διαπραγματεύσεων, ενώ υπήρξε μια κλιμάκωση των βιοπραγιών που στόχο είχε να παρεμποδίσει την ειρηνευτική διαδικασία των Μαχάσετ στην οποία συμμετείχαμε όλοι. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτή θα καταλήξει σε μια πολιτική λύση για την Μαροκινή Σαχάρα. Και το Μαρόκο θέλει μια τέτοια πολιτική διαπραγμάτευση. Εγώ δεν επρόκειτο να θέξω αυτό το θέμα, αλλά με προκαλέσατε. Πόσα λεπτά έχω ακόμη. Έπρεπε να είχατε ήδη τελειώσει. Μάλιστα. Αυτή η αποστολή των 7 μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Μαρόκο δεν είχε καμία οικογενειακή απόχρωση. Ουσιαστικά ήθελαν να επιδιώξουν κάποιους πολιτικούς στόχους στη συνεργασία με τις ε, εξωτερικές ε, υπηρεσίε πληροφοριών. Το Μαρόκο δεν έχει κανένα κόμπλεξ ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για, την, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κανείς δεν με ρώτησε εδώ, γιατί πρόσφατα ο Αλγερινός Υπουργός όταν ερωτήθηκε για τους Σαχαραουίτες στο Τιντούφ, δεν απάντησε. Δεν έδωσε καμία απάντηση. Εκείνη που υπάρχει πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Αλγερινή Σαχάρα και όχι στη Μαροκινή. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάννη και Γραμματεύ. Παρακαλώ τον επικεφαλής αντικοσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ενίκο Λανταμπούρου, να είναι όσο πιο συνοπτικός γίνεται, διότι ο Υπουργό ο κ. Μπουγκάιτ ε, περιμένει έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικά λεπτά. Έχουμε και τα συμπεράσματα επίση. Juste pour répondre à Madame Για να απαντήσω στην κυρία Φλότ στο τελευταίο της ερώτημα, θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει αυτό που με ρωτά αν υπάρχουν κριτήρια για να κρίνουμε το δημοκρατικό καθεστώ μια χώρα, για να μπορεί να μπει στο ενισχυμένο καθεστώ, Όχι, δεν υπάρχουν κριτήρια τη Κοπενχάγη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κατά την άποψή μου είναι έξοχο το ερώτημα που μπροστά στην αοριστολογία την καλλιτεχνική που έχουμε μπροστά μας και για να μπορέσουμε να καλύψουμε και άλλες χώρες αυτό το καθεστώς, αν δεν καθορίσουμε κριτήρια και, και κινούμε θα κατά περίπτωση θα ξεφύγουμε κάπου από το δρόμο μας. Άλλο ερώτημα, τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο για να ελέγξει τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις και την πρόοδο όσον αφορά το καθεστώς. Συνεχίσει, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει ε, είναι το καλύτερο. Υπάρχουν έγγραφα κυρία μου ετήσια έκθεση για την πολιτική γειτονία, χάρη, ετήσια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσεω για το Μαρόκο. Υπάρχουν εκθέσει που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποστέλει στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει πληροφορίε από αυτόν. Επόμενη Δευτέρα γίνεται σημαντική συνεδρίαση, ετήσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνδέσεως με το Μαρόκο για τη Συμφωνία σύνδεση Σε αυτό το Συμβούλιο θα γίνει απολογισμός του πρώτου έτους ε, του ενισχυμένου καθεστώτος. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί εγγράφου που έχει κάποιο ενδιαφέρον που θα μπορούσε να συζητηθεί ε, με τους βουλευτές στην Ολομέλεια ή διμερός σε οποιοδήποτε σχήμα. Εγώ πιστεύω ότι η σε Επιτροπή εφαρμόζει μεγάλη διαφάνεια από αυτόν. Από εσά εξαρτώνται οι πρωτοβουλίε για να ζητήσετε την εκτελεκτική εξουσία ε, να σα έρθει να σα ενημερώσει. Εγώ που ήμουν νέο, όταν ήμουν νέος συμβουλευτή, ξέρω τι είναι η πτύψη αυτή για ανάλυση και για πληροφορίε ε, για να κάνει τη δουλειά του ο βουλευτής. Άλλο ερώτημα που ετέθη, αν πρόκειται περί μοντέλου αυτό το ενισχυμένο, ενισχυμένο καθεστώς. Όχι, είναι ένας πειραματισμός πολιτικός θα έλεγα. Καταλαβαίνω ότι οι ακαδημαϊκοί που έχω δίπλα μου αρέσκονται στο να φτιάχνουν οι δυτικές πράξεις και να εξετάζουν τα θέματα συνθήκων κλπ. Ε, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά εδώ που βρισκόμαστε. Θυμάμαι ότι με τον πρόεδρο πρώτη τα ξεκίνησε η ιδέα της πολιτικής γειτονίας όταν τελειώναμε τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις νέες χώρες. Φτιάχναμε το μονοπάτι προχωρώντας. Βλέπαμε και κάναμε. Βέβαια δεν είναι ικανοποιητικό, πρέπει να καθοριστούν κάποια κριτήρια όπως αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως όσον αφορά τα κριτήρια περί δημοκρατίας κλπ. Αλλά το ενισχυμένο καθεστώς αντι αντιστοιχεί σε μια ιδιαίτερη κατάσταση που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Μαρόκο και τη βούληση της χώρας όπως προανέφερα να έχει σαφή στρατηγική προσέγγιση. Από εκεί μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν είναι ένα μοντέλο, είναι πειραματισμός πολιτικός χωρίς να έχει σαν στόχο προσχώρηση για προσέγγιση στο μέγιστο δυνατόν μεταξύ συμφωνίας, κάτι μεταξύ συμφωνία σύνδεση και προσχώρησης είναι. Μπορούμε να συζητήσουμε πολιτικά τι γίνεται. Δεν θέλουμε όμω να επικρατεί παντού συνοχή, διότι η Αίγυπτος δεν είναι Μαρόκο, η Λιβύη ακόμα λιγότερο κλπ. κλπ. Στη μεσογειακή πολιτική σήμερα έχουμε ένα επίπεδο ε, που δεν λειτουργεί, ε, που τη Ένωση για το Μαγκρέ που δεν λειτουργεί. Έχουμε διμερεί επαφέ με κάθε μία από τι χώρε αυτέ που θέλουν συναρτήσει των φιλοδοξιών του έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν. Με μεγάλε διαφορέ. Αν το Ισραήλ έχει προχωρήσει κάποια πράγματα, τι να πω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα πρέπει να καθυστερεί το Μαρόκο λόγω του Ισραήλ και κανένα άλλο. Κατά περίπτωση μπορούμε να δούμε τι πρέπει να γίνει πριν να κάνουμε μεγάλα ε, σχέδια, γενικά σχέδια και να προσπαθούμε να καθορίσουμε διάφορα πράγματα. Η Ένωση για το Μαγκρέμπ είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ότι πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία ανακοίνωση για την κατάσταση στο Μαγκρέμπ και τις αναπτυξιακές δυνατότητές του. Και η τότε Προεδρία δεν έθεσε ως προτεραιότητα στο πρόγραμμά της αυτό το θέμα. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια αμφιβολία, δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί να κάνει κάτι. Θέλει να προωθήσει τα πράγματα, αλλά θα πρέπει και οι διάφοροι και τα κράτη-μέλη να δώσουν μια όθηση ώστε να έρθουν τα εμπόδια στην Ένωση του Μαγκρέπ. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, υπάρχει ένα σχέδιο, μαρακινό σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας που χαίρει της ευρωπαϊκής υποστήριξης προσπαθεί το σχέδιο αυτό να μειώσει την κατανάλωση, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει ενάβσματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διευρύνει, να διαφοροποιήσει τις πηγές ανεφοδιασμού, τους προμηθευτές. Και εμείς αντίστοιχα προβλήματα έχουμε με το Μαρόκο, γιατί ούτε και το Μαρόκο έχει ορυκτό πλούτο. τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα υπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την ενεργειακή πολιτική, ώστε να μπορέσουν και τα μεγαλύτερα δίκτυα ενέργειας από την Νότια Αφρική να διέρχονται από το Μαρόκο και να τροφοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ήδη υποσυζήτηση αυτό το θέμα και κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε. Μιλήσατε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τέθηκε μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον κύριο Γκουράκη. Το Μαρόκο. Για το Μαρόκο, μάλλον η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, να ζητούν από τις, Ευρωπαϊκές, από τις Μαροκινές Αρχές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών με τον Ευρωπαίο Πρέσβη σε τακτικές ε, συναντήσεις όπου γίνονται ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών για το τι συμβαίνει στο Μαρόκο και το κατά πόσο υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε ζητούμε αν χρειαστεί εξηγήσει από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, χρηματοδοτούμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεκδικούν την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής δημοκρατίας. Έχει καταθάσει ο Υπουργός Εξωτερικών του, της Αιγύπτου. Τώρα, είμαστε παρατηρητές στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο γραφείο μας και θα σας δώσουμε πιο λεπτομεριακές πληροφορίες για το τι κάνουμε. Ξέρετε ποια είναι η δέσμευση και προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ανθρώπινα δικαιώματα και το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο γιατί αποτελεί σήμα κατά τεθέν της εξωτερικής μας πολιτικής και αυτό το γνωρίζει και η κυβέρνηση του Μαρόκου γιατί συχνά είμαστε πολύ φορτικοί σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση πληροφοριών από το Μαρόκο. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υποστηρίζει απερίφραστα και ανενδίαστα τις ε, προσπάθειες του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέως και του εκπροσώπου του στην ε, προσπάθεια ειρηνευτικής διαδικασίας, προκειμένου να διαθετηθεί το θέμα. Όταν ήμουν μάλιστα στις Βρυξέλλες, δεχόμουν ε, εκπροσώπους του μετόπου Πολυσάριο είχαμε τακτικές επαφές με τις μαροκινές αρχές. Χρειαζόμαστε μια πολιτική λύση που περνάει από τη διαπραγμάτευση στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτή την ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγύδα του ΙΕ υποστηρίζουμε. Φυσικά κάποια κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ευαισθησίες και άλλες θέσεις, αλλά αυτή είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ένωσης. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λανταμπούρου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μου. Ο φίλο μα, ο κ. Αντώνη Παντσιέρη, επικεφαλή αντιπροσωπεία για τι σχέσει με το Μαγκρέμπ και με την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, έχει το λόγο. Εφόσον υπάρχει ήδη εδώ Αιγύπτιο Υπουργό, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ συνοπτικό. Θα είμαι τάχιστο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προφανώ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τον πρόεδρο αυτή για τη δυνατότητα που μα έδωσε. Συζητήσαμε ευρέω, πιστεύω, σήμερα με του τρει συγητέ στον καινοτόμο χαρακτήρα του κοινού αυτού εγγράφου θα ήθελα να υπογραμμίσω μια πτυχή του λόγω εγγράφου, δηλαδή ότι εμείς καθιστούμε επιτέλους δυνατή τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής μικτής και αυτό επιτρέπει πλέρα από το χρόνο που δεν υπάρχει να μιλούμε με ειλικρίνεια σε αυτή την επιτροπή και για θέματα τα οποία θίγησαν εδώ και χαιρετίζουμε το, ενισχυμένο αυτό καθεστώς. Είναι μετριοπαθής φορέας Απαραίτητο φορέας στο Μαγκρέμπ το Μαρόκο και βοηθά να εφαρμόσουμε τι δεσμεύσει που αναλάβαμε όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, την πολιτική γειτονία. Ενισχύεται η ολοκλήρωση, δίνει αποτελέσματα αυτή η πολιτική. Στην επαφή με τον ευρωπαϊκό χώρο και δημιουργεί μεγαλύτερο κοινωνικό και ε, οικονομικό χώρο. Δεν θα σταθώ σε αυτό, διότι ευρέω ε, ανελήθη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μόνο δύο πτυχέ εν τέλει πολιτικός ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Σαμράνη αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα και υπογράμμισε πως το Βασίλειο του Μαρόκο δημιούργησε μηχανισμό στενότητα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κόσμο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχουν πιο σαφεί δεσμεύσει όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα ήταν χρήσιμο, διότι υπενθυμίζω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων, τα θέματα τη ελευθερία για μα είναι ε, στο επίκεντρο και μάλιστα σήμερα που έχει τεθεί σε ισχύ το, η συνθήκη της Λισαβόνα. Θα ήταν χρήσιμο στην ανάπτυξη αυτού του καθεστώτος να υπάρξει επαρκής κάλυψη, επαρκής χώρος για αυτά τα θέματα. Και μπορούμε με δύο τρόπους να το πετύχουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα να προβλέπουμε και πολιτικές ελέγχου, εποπτείας όσον αφορά το θέμα και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο αυτό είναι το αίτημα που θα πρέπει να προωθηθεί και είναι δίκαιο. Και το άλλο είναι να συμμετάσχουν οι οργανωμένε ε, μορφέ τη κοινωνία των πολιτών. Δεν θα πρέπει να φοβούμε τη συζήτηση και το διάλογο. Δημιουργούμε μια διαδικασία ενισχύσεω των σχέσεων και πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία ενισχύσεω των σχέσεων πρέπει να δημιουργήσει προποθέσει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική ολοκλήρωση αλλά και δημοκρατική ολοκλήρωση των χωρών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε για, αυτή την, ε, για αυτό το αποτέλεσμα και θα πρέπει όλοι οι βουλευτές να μπορούν να συμβάλλουν ε, της μεικτής ε, επιτροπής που θα δημιουργηθεί ε, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους το ταχύτερο δυνατόν. Και ο καθηγητής Μάρτιν αναφέρθηκε σε κάποιες αντιφάσεις που υπάρχουν όσον αφορά τα διάφορα προθυμένα καθεστώτα και πώς διαφέρουν μεταξύ τους. Θα πρέπει να εργαστούμε σοβαρά για να πετύχουμε τον προαναφερθήτα στόχο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ όσους πήραν το λόγο, ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και παραγωγική. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερή διάταξη με τα δύο λεπτά διαλύματο που είναι αναγκαία για να αλλάξουμε θέσει. Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με κάποια καθυστέρηση την ε, ακρόασή μας με τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τον κύριο Αχμέτ Αμπούλ Γκέιτ. Ενώ εσείς καθόσαστε και εφόσον δεν έχει... Θα ήθελα να πω ότι η ανταλλαγή απόψεων με Μαρία Τρεσάκε για την ad hoc αντιπροσωπή 14-16 ε, Νοεμβρίου την αντιπροσωπή στο Κωσυφοπέδιο δεν μπορεί να γίνει σήμερα αυτή η ανταλλαγή απόψεων διότι περάσαμε ε, λόγω των προηγούμενων συνομιλιών το χρονικό περιθώριο και θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση αυτή στα πλαίσια του διευρυμένου Προεδρίου για να θέσουμε το θέμα αυτό που αφορά την ακρόαση με τον είπα εκπρόσωπο. Μου είπε ανταλλαγή απόψεων, μου λέει ο συνάδελφο. Ανταλλαγή απόψεων με τον ήπατο εκπρόσωπο τη Ενώσεω. Με την ήπατη Ύπατη εκπρόσωπο. Μπορούμε τώρα λοιπόν να περάσουμε στην έναρξη των εργασιών μας, καλωσορίζοντας τον κύριο Υπουργό, που μαζί με τους συναδέλφους της αντιπροσωπείας ε, είναι εδώ με τους εκπροσώπους αντιπροσωπείας σε σχέση με το Μασρέκ. Και να πω δύο πράγματα. Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος νομίζω από την προηγούμενη επίσκεψη του Υπουργού στο Κοινοβούλιο και αυτό έχει μια σημασία όχι τόσο συμβολική αλλά δείχνει θα έλεγα τη σημασία που δίνουμε δείχνει εμπράγματα τη σημασία που δίνουμε στο διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει η χώρα σας ε, ε, στον περίπλοκο χώρο της Μέσης Ανατολής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις ε, εξελίξεις στην περιοχή σας και γι' αυτό εμπνευστήκαμε σε αυτή την Επιτροπή να ξαναδημιουργήσουμε την ομάδα εργασίας για τη Μέση Ανατολή, της οποίας προείδρευε ο φίλος ο κύριος Hans Gerd Πίτερινγκ και συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να ξέρουμε κύριε Υπουργέ ποια είναι η άποψή σας για την ειρηνευτική διαδικασία και για την διαμεσολάβηση της χώρας σας όσον αφορά το θέμα της Παλαιστίνης. Έχουν δημιουργηθεί αβεβαιότητες όσον αφορά το πολιτικό προσκήνιο στη Μέση Ανατολή ο κύριος Μαχούντα Μπάς, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, διαπραγματεύτηκε με ισορροπημένο τρόπο αυτές, αυτές τις σχέσεις ε, αποφάσισε να μην υποψήφιο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και δεν γνωρίζουμε ε, πότε θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές. Είναι καλό ότι ανακοινώθηκε ένα πάγωμα όσον αφορά τους επικισμούς τους Ισραηλινούς αλλά μειώνεται αυτό το θετικό μέτρο διότι είναι προσωρινό μέτρο που ανακοινώθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Όμως εξαιρείται η Ιερουσαλήμ, η Ανατολική Ιερουσαλήμ από αυτό το μέτρο. Ταυτόχρονα μία επίλυση της συγκρούσεως που βασίζεται στη δημιουργία δύο κυρίαρχων κρατών είναι κάτι που χρειάζεται κατεπηγόντως να υλοποιηθεί και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει πολύ την ε, μεσογειακή μας ε, εταιρική σχέση η, η ακύρωση της συνεδριώσεως των Υπουργών Εξωτερικών για τη Μεσογειακή Ένωση είναι κάτι που το αποδεικνύει. Συμπροεδρεύει η χώρα σας της Ενώσεως για τη Μεσόγειο και γι' αυτό και αυτό είναι ένας λόγος να ζητήσουμε κύριε, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ να σχολιάσετε τις πολυμερείς σχέσεις στην, ε, των χωρών της Μέσης Ανατολής. Σας δίνω παρεφή το λόγο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρόνο που θεωρείτε απαραίτητο, αλλά καλό θα ήταν αν μιλήσουμε εμεί λιγότερο να αφήσουμε περισσότερο να μιλήσουν συνάδελφοι. Έτσι θα έχετε περισσότερο χρόνο να δώσετε και απαντήσει. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Thank you. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία αυτή για μένα να επανέλθω. Δύο φορές έχω έρθει μέσα σε 12 μήνες να μιλήσω σε αυτήν την Επιτροπή. Και αυτό το γεγονός δείχνει τη μεγάλη δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μου η Αίγυπτος για την ενίσχυση και εδραίωση των σχέσεών μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν πρέπει να πω ότι πράγματι προέρχομαι από μία περιφέρεια Δεν θέλω να πω μια προβληματική περιφέρεια, αλλά προέρχομαι από μια περιφέρεια η οποία ναι μεν έχει δυσκολίες και προβλήματα αλλά προσπαθεί αυτά να τα ξεπεράσει. Όπως πολύ σωστά τονίσατε έχουμε το πρόβλημα το Μέσο Ανατολικό, την Παλαιστινιακή Ισραηλινή διένευξη, την Άραβο Ισραηλινή διένευξη είναι πολλαπλές πτυχές ενός προβλήματος που βασανίζουν την περιοχή μας. Έχουμε όμως και το θέμα μιας χώρας όπως το Σουδάν που έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε το κέρα της Αφρικής ε, με όλα τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από εκεί. Έχουμε τη Σομαλία, το πρόβλημα της πειρατείας, ε, το πρόβλημα του χάους που επικρατεί στην περιοχή εκεί. Έχουμε βεβαίως ε, την Μεσογειακή Ένωση η οποία άρχισε, εγγενιάστηκε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2008 και από τότε έχει μείνει στάσιμη αυτή η Ένωση. Ε, παρόλο που τομεακές ε, υπουργικές συναντήσεις γίνονται. Όμως, η Μεσογειακή Ένωση ε, και η γραμματεία της θα πρέπει να εξασφαλίσει την εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν γίνει. Είναι λοιπόν μια περιοχή του κόσμου πάρα πολύ σημαντική για την παγκόσμια σταθερότητα, δεδομένου ότι 60% των ενεργειακών πόρων όλης της υφηλίου ε, προέρχονται από αυτή την περιοχή, ε, την Αραβική Χερσόνησο, τον ε, Αραβικό κόλπο και σε αυτή την περιοχή έχουν προκύψει εκ νέου εντάσεις μεταξύ του Ιράν και των χωρών της Δύσης. Δεν θα έλεγα χώρες της Δύσης, αλλά θα έλεγα τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένης τώρα και της Γερμανίας. Άρα λοιπόν αυτή η περιοχή του κόσμου πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι μία περιοχή η οποία θέλει να αναπτυχθεί, θέλει να αναπτυχθεί στο, στα, σε επίπεδα του προηγμένου κόσμου, αλλά είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν φοβερές επιπτώσεις στους ε, πληθυσμούς αυτής της περιοχής. Θα απαντήσω με μεγάλη χαρά στις ερωτήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων, εδώ στο σώμα είτε αφορούν τον Παλαιστινιακό-Ισραηλινό διάλογο είτε τις Ισρα... Παλαιστινιακές Ισραηλι... Ισραηλινές ε, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις είτε τον διάλογο με την Αίγυπτο, Αίγυπτο-Ισραήλ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στη συνάδελφο, στη κυρία Ρίζα Ματίας που εκπροσωπεί το πρόεδρο Μάριο Νταβίντ, τον πρόεδρο της ε, κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για το ΜΑΣΡΕΚ. Σας ευχαριστώ. Όπως είπατε, αναπληρώνω τον Μάριο Νταβίντ, που είναι ο πρόεδρος της ε, κοινοβουλευτικής αυτής αντιπροσωπείας και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λισαβόνα στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη θέση ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίαση που μας έκανε και για την σύντομη εισαγωγή που μας έκανε και που δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να προβούμε σε μια διεξοδική ανάλυση της κατάστασης της περιοχής και οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή αυτή είναι τεράστιες, ε, κάτι που συνειδητοποιούν όσοι την επισκέπτονται. Είχαμε πολλές σχέσεις με τις ε, Αιγυπτιακές ε, αρχές και μέσω της ε, Επιτροπής μας ΡΕΚ. Είχαμε και τακτικές επισκέψεις ε, και τις αντιπροσωπείες μας ε, στην Αίγυπτο και δικός εκπροσώπος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατα είχαμε αποστολή της αντιπροσωπείας μας στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Και μάλιστα η έκθεση πεπραγμένων αυτής της αποστολής βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας για όποιον ενδιαφέρεται. Δεν μπορούμε τώρα να αναλύσουμε το σχέδιο επαφών που είχαμε με τις Αιγυπτιακές Αρχές. Καλύτερα να αφιερώσουμε το χρόνο που έχουμε στις ε, ερωταπαντήσεις, ώστε να ικανοποιηθούν οι απορίες των Ευρωβουλευτών και να έχουμε έναν γόνιμο διάλογο για όλα τα θέματα που ανέφερε ο Υπουργός ή τα θέματα που ενδεχομένω θα θέξετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Ζήτησε το λόγο ο κ. Σαλαφράγκα, που μπορεί να μιλήσει. Παρακαλώ δύο λεπτά αν έχετε την καλοσύνη μόνο. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό και να εκφράσω την ιδιαίτερη μου εκτίμηση για την προθυμία και τη διαθεσιμότητά του για την ανταλλαγή απόψεων ε, μαζί μας, γιατί και η αναπληρώτρια του Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας μας, ΡΕΚ, μίλησε για, τις, μίλησε για τις τακτικές επαφές ε, που είχατε και μάλιστα είχατε συνάντηση και με τον Πρόεδρο Πέτερινγκ, ε, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε διμερεί σχέσει πολύ πλούσιε. Είμαστε ο πρώτος εμπορικός εταίρος στη χώρα σας και ο δεύτερος επενδυτής στην Αίγυπτο μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και μάλιστα ο ρόλος που διαδραματίζει η Αίγυπτος στο Μεσανατολικό είναι πολύ σημαντικός. Ερωτώ λοιπόν κύριε Υπουργέ, πώς βλέπετε τη δέσμευση της νέας Αμερικανικής ε, κυβέρνησης ε, στη διαμάχη αυτή. Γιατί το είπαμε και στο Στρασβούργο, στην ομάδα εργασίας που ε, στην οποία προεδρεύει ο κύριος Πέτερινγκ. Πώς βλέπετε την κατάσταση του μεσανατολικού ζητήματος και πού οφείλεται η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων ή σε τι εμπόδια προσκρούει η επανάληψη των συζητήσεων. Χαίρομαι που μετά τις δυσκολίες έχουμε κάποια συσπήρωση πάλι της Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας και θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, σε μία μεταβατική στάση της οικονομίας σας πώς επηρεάζεστε από την χρηματοπιστωτική κρίση και πώς βλέπετε τη συμμετοχή της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα και γιατί σεβαστήκατε το χρόνο που σας διατέθη. Ο κύριος Ομπιόλς για δύο λεπτά. Ε, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για την Ένωση για τη Μεσόγειο και διαπιστώσατε κάτι που είναι προφανές την ύπαρξη κάποιας αποτελμάτωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι πολλοί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση με αμηχανία και μεγάλη ανησυχία. Έχουμε την αίσθηση ότι το σχέδιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο στην οποία συμπροεδρεύει ο πρόεδρος της χώρας σας μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ε, θα σηματοδοτούσε τη μετάβαση σε μια πιο συγκεκριμένη φάση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ε, της ε, Νότιας και Ανατολικής Μεσογειακής Λεκάνης. Ήταν μια ένωση σχεδίων, όπως δήλωνε ο πρόεδρος Σαρκοζή. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια πιο ευάλωτη ε, δομή από ό,τι φαινόταν. Φαίνεται ότι γίνεται έρμεο της ε, ε, Ισραηλοπαλαιστινιακής διαμάχης και δεν στηρίχθηκε αρκετά στην πολυμερή διαδικασία της Βαρκελόνης που άντεχε περισσότερο στις αλλαγές της συγκυρίας και ήταν και πιο ανθεκτική στην κρίση. Αναβλήθηκαν ε, ε, τα Υπουργικά Συμβούλια στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρθηκατε και στις άτυπες υπουργικές ε, συζητήσεις που είτε αναβλήθηκαν ήταν πολύ δυσχερής η διεξαγωγή τους. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια όθηση στην Ένωση για τη Μεσόγειο και θα ήθελα και μια διευκρίνηση για το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την κατάσταση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ένα κρίσιμο πρόβλημα ποια θα είναι η σχέση που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της ε, ανάπτυξης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και των εξελίξεων στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή διένεξη. Και μάλιστα πιστεύετε ότι η αποτελμάτωση της Ένωσης για τη Μεσόγειο οφείλεται στην αποτελμάτωση του Μεσανατολικού ή πιστεύετε ότι η καλύτερη όθηση για την ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού είναι μία προώθηση της ε, κατάστασης στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ κύριε Αμπιόλς. Νέιτς, το επόμενο όνομα για δύο λεπτά. Κυρία Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρέσβυρα, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται. Θα προσπαθήσω να, υπογραμμίσω την Παλαιστινιακή κρίση να αναφερθώ σε αυτό το θέμα και από τη μία πλευρά υπάρχει η Παλαιστινιακή Αρχή στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και από την άλλη πλευρά η Αμάς στη Γάζα. Ξέρουμε ότι η Αίγυπτος κάνει ό,τι μπορεί. Προσπαθεί να συμβάλλει σε μια συμφιλίωση. Ίσως μεγάλη λέξη είναι αυτή, μεγάλη κουβέντα, αλλά συνεννόηση μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Μπορείτε να μας πείτε αν βλέπετε προπτική, λύσεις ή θεωρείτε ότι αντιθέτως ότι τα δύο στατόπεδα, το τα δύο παλαιστινιακά στατόπεδα, αν μπορώ να το πω έτσι, σκληραίνουν τη θέση τους, εμποδίζοντας έτσι, πιστεύω, κάθε ουσιαστική πρόοδο για την επίλυση του προβλήματος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Έχοντας γίνει κάπως κοινική πλέον μπορούμε να πούμε ποιον, σε ποιον είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Το ότι η Παλαιστινιακή Αρχή από τη μια πλευρά και η Χαμάς από την άλλη δεν συνεννοούνται ή δεν καταφέρνουν να βρουν ένα ελάχιστο παρονομαστή συνεννόησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νάιτς. Πουέρτα για δύο λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου που είχε την καλοσύνη έρθει στη συνεδρίασή μας. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. η πρόσφατη, το πρόσφατο δημοψήφισμα στην Ελβετία για τα τζαμιά, πώς, τι απήχηση είχε στην Αίγυπτο. Δημιουργήθηκαν κάποιες ανησυχίες. Ποια ήταν η αντίδραση που προκάλεσε στην Αίγυπτο η έκβαση αυτού του δημοψηφίσματος στην, ε, στην Ελβετία. Έχω και μία ερώτηση για την Ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση. Υπάρχει μια αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ίδια πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή για μια ε, επαναφορά στην Τράπεζα των Ειρηνευτικών Διαπραγματεύσεων. Η Αίγυπτος είναι ένας προνομιούχος εταίρος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτώ λοιπόν, όχι τι έκανε η Αίγυπτος για να βρεθεί μια πολιτική λύση με βάση ξεκάθαρες αρχές για το Ισραήλο-Παλαιστινιακό, αλλά σας ερωτώ τι έκανε η Αίγυπτος στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαδραματίσει ένα σαφέστερο ρόλο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού εντός ε, του Αιγυπτιακού κράτους. Ευχαριστώ κύριε Πόρτα. Ο κύριος Πέτερινγκ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα ξανά τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και κύριε Υπουργέ, πρέπει να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή της Αιγύπτου στην ενευτική διαδικασία στην ε, περιοχή της ε, Εγγύς Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και προϋποθέτει έντονη πολιτική βούληση και αυτό το αναγνωρίζουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Εμείς στην Ευρώπη, το είπα και χτες στους καλεσμένους μας, δεν θα επιτρέψουμε την υπονόμευση της ασφάλειας του Ισραήλ. Και όταν από τον ε, πρόεδρο του Ιράν ακούμε ότι θα πρέπει να ε, σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη του κόσμου και όταν ακούμε αυτές τις ε, δηλώσεις ομολογώ ότι τις θεωρούμε απαράδεκτες. Απαράδεκτο όμως επίσης είναι το γεγονός να επεκτείνει ε, το, το, το ε, χτίσιμο κατοικιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ και σε άλλες περιοχές διότι ποτέ δεν θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα αυτό και ποτέ δεν θα ζήσουν σε ειρήνη το Ισραήλ και η Παλαιστίνη αν συνεχιστούν αυτές οι προκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ε, αν πιστεύετε ότι θα πρέπει ο, τα Ηνωμένα Έθνη να ασχοληθούν εκ νέου με την νέα επεκτατική ε, πολιτική ε, του Ισραήλ για την επέκταση του χτισήματος των κατοικιών. Ευχαριστώ κύριε Πέτερινγκ. Για δύο λεπτά η κυρία Μούνιτς έχει το λόγο. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα και εγώ να ασθενιστώ τις ανησυχίες των προλαλισσάντων για την Ένωση για τη Μεσόγειο, στην οποία συμπροεδρεύει η Αίγυπτος. Ποιες είναι οι προοπτικές για να αρχίσει να λειτουργεί η γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η Αίγυπτος ε, εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύσφυξη και βάθηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εδραίωση της δημοκρατίας και οι εμπορικές συναλλαγές. Υπάρχουν όμως προοπτικές για να αποκτήσει και η Αίγυπτος ένα ενισχυμένο καθεστώς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει και το Μαρόκο. Ποιες είναι οι αιγυπτιακές προοπτικές ό,τι αφορά το, την πιθανότητα σύναψης εγγράφου ενισχυμένου καθεστώτος. Σας ευχαριστώ κυρία Μόνιτς, Βάιγκλ για δύο λεπτά. Ο κύριος Βάιγκλ. Ε, Spoštovani gospod minister, ενότνοστ palestincev η έλλειψη ενότητας μεταξύ των πολυστηλίων μας ανησυχεί πολύ και εσάς βεβαίως. Εσείς όπως κανείς άλλος έχετε την καλύτερη δυνατότητα να εργαστείτε για την εξέβρεση μιας λύσης. Αυτή η έλλειψη ενότητας όμως αποτελεί και μία δικαιολογία της πολιτικής του Ισραήλ, η οποία βασίζεται επί των κεκτημένων δικαιωμάτων. Είναι ένα προπέτασμα καπνού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι ρόλο νομίζετε ότι μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δει τώρα που ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία μας δίνει περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερη δύναμη ε, για το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρετε ποια είναι η άποψή σας για την ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ και έλαν για δύο λεπτά. Έχει το λόγο. Κύριο Κύριε Υπουργέ, εκτιμώ το ρόλο της Ευρώπης ε, στην ε, συμβολή ως κράτος το οποίο συμβάλλει στην ειρήνη της ε, λεκάνης της Μεσογείου. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα για την δέσμευση της ε, Αιγυπτιακής διπλωματίας να επιτύχει ρεαλιστικούς στόχους και να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη. Όλοι βεβαίως ανησυχούμε για την παρούσα κατάσταση. Η Αιγύπτ η Αίγυπτος ε, έχει ένα σημείο, ε, ένα πέρασμα με την λωρίδα της Γάζας η, η, πώς μπορεί λοιπόν η Αιγυπτός να ε, συμβάλλει στην άμβλυνση της ανθρωπιστικής, του ανθρωπιστικού προβλήματος στην Γάζα και να διασπάσει αυτή την απομόνωση της λωρίδας της Γάζας από τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Κέλαμ. Ράουτσεκ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Κύριος Ράουτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, για το Αφγανιστάν ο Αμερικανός πρόεδρος ε, θα ανακοινώσει πολύ σύντομα την αύξηση των Αμερικανικών δυνάμων. Οι Βρετανοί συνάδελφοι επίσης έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν 500 περισσότερους στρατιώτες, στρατιωτική δύναμη. Ποια είναι η γνώμη σας για το Αφγανιστάν και για την περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας. Να αυξηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε μια ικανοποιητική μεσοπρόθεσμη πολιτική, υπάρχει μια ε, ικανοποιητική πολιτική εξόδου των στρατιωτικών δυνάμεων, απόσυρσης, τι πιστεύετε. Ευχαριστώ. Παρβάνοβα, η κυρία Παρβάνοβα, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις ένας από τους παίκτες κλειδιά στην περιφέρεια αυτή είναι το Ιράν. Συνεχώς υπάρχουν, ακούμε, ε, πλοία να να, με, με, όπλα, ε, φορτωμένα με όπλα, ε, τα οποία προορίζονται για τους Χεσμολά και το Ιράν διαψεύδει την αποστολή οπλισμού προς την οργάνωση αυτή. Ποια είναι η άποψή σας. Και δεύτερον, Πρόσφατα ανακοινώθηκε από Ιρανούς αξιωματούχους ότι προ... προτίθενται να χτίσουν, να κατασκευάσουν πέντε ακόμα πυρηνικά εργοστάσια. Ποια είναι η γνώμη σας και σε αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Γκουαλτιέρη, για δύο λεπτά. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Στην παρέμβασή σας αναφερθήκατε και στο κέρας της Αφρικής και στη Σομαλία περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποστολή, την αποστολή Αταλάντη. Υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την προσπάθεια και ότι θα πρέπει, είπαμε, να αντιμετωπιστούν και τα αίτια της πειρατείας. Και γι' αυτό και η αποστολή που προβλέπεται, που γραμμάζεται της ΚΕΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην ε, Σομαλία. Πώς βλέπετε εσείς τη διαδικασία του Τζιμπουτή, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα στην Αφρικανική Ένωση, όχι μόνο υποστηρίζοντας την μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά μέσω της ενίσχυσης περιφερειακής προσέγγισης στην κρίση της Σομαλίας. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Κλείνουν οι παρεμβάσεις με τον συνάδελφο Τάκουλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό το εξής. Η Αίγυπτος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι μπορεί να κάνει η Αίγυπτος για να υποχρεώσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τον Ισραηλινό στρατιώτη. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τη βοήθεια της Αιγύπτου και μπορεί να παίξει ένα πραγματικό ρόλο στην απελευθέρωση αυτού του στρατιώτη. Σας ευχαριστώ κύριε Τάκουλα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Υπουργό που έχει χρόνο να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Αν αυτές είναι όλες οι ερωτήσεις που θέλετε να απαντήσω, ευχαρίστω να τις απαντήσω και να είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω από την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η άποψή μας για την νέα αμερικανική κυβέρνηση και την, τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσει. Πιστεύω ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει όλη την καλή θέληση να κάνει κάτι, να επέμβει. Και πιστεύω ότι η πρώτη μέρα του νέου πρόεδρου της Αμερικής, όταν εχρήστη πρόεδρος, την επόμενη μέρα ε, στο Λευκό Οίκο όρισε τον ε, γερουσιαστή George Mitchell ως ειδικό εκπρόσωπο ε, της περιοχής μας. Αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ε, ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες βασιζόμενοι σε μία κατανόηση, σε μία συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ενωμένων Πολιτειών. Ζήτη λοιπόν από το Ισραήλ να σταματήσει κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και, και στη δυτική, συγγνώμη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και προσπαθεί να λάβει ορισμένα βήματα προς τους Ισραηλινούς για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η δική μας τάση είναι προς την Αμερικανική κυβέρνηση. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε την πολιτική σας υπό αυτή τη γωνία, εντάξει, οκ, θα σας υποστηρίξουμε. Όμως, η θέση της Αιγύπτου ήταν πάντοτε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο τέλος, στην τελική φάση του, της υπόθεσης, δηλαδή πώς το, η τετράδα ε, Ηνωμένε Πολιτείε, Ευρώπη, Ρωσία και Ισραήλ θα μπορέσουν να ορίσουν το τελικό πλαίσιο της επίλυσης του προβλήματος και, και δει πώς θα ορίσουν τα σύνορα του Παλαιστινιακού κράτους. Εάν λοιπόν το τελικό βήμα προϋποθέτει την εδραίωση, τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βήμα που είναι ο καθαρισμός των συνόρων αυτών που κάποια στιγμή θέλουμε να δημιουργηθούν. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για περιοχές που έχουν καταληφθεί από το 67. Όμως, αυτά τα εδάφη, αυτά τα εδάφη είναι ίσα σε έκταση με τα εδάφη τα οποία κατελήφθησαν τον Ιούνιο του 67. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι έχουν χάσει από, στους Ισραηλινούς 2.600 τετραγωνικά 2.660 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οπότε θα έπρεπε το Ισραήλ να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να έχουν έλεγχο σε μια αντίστοιχη ισότιμη εδαφική έκταση. και θα ελέγχει το Ισραήλ, ό,τι είναι μέσα στα σύνορά του θα είναι εδάφη του Ισραήλ και ό,τι είναι μέσα στα σύνορα της Παλαιστίνης θα είναι εδάφη των Παλαιστινίων. Αυτή ήταν η στάση μας. Σήμερα έχουμε μία δήλωση από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να εφαρμόσει ένα μορατόριο στην Δυτική Όχθη και δυστυχώς το ανέφερε την περιοχή αυτή ως Ιουδαία και Σαμάρια. Άμα, άμα, άμα μιλάς περί Ιουδαίας, τότε δεν είναι δυνατό να την αναγνωρίσεις αυτή την περιοχή ως ε, Παλαιστινιακή έπρεπε να πει δυτική όχθη, ζητική όχθη και να πει ότι θα σταματήσουμε να χτίζουμε οικισμούς στη δυτική όχθη. Διότι αν πει Σαμάρια και Ιουδαία, πώς είναι δυνατόν τότε να δώσεις τα εδάφια αυτά στους Παλαιστινίους, ε, αφού εξορισμού δεν θα είναι δικά τους, άμα τα περιγράφεις με αυτή την ορολογία. Δεύτερον, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι η Ιερουσαλήμ είναι κυρίαρχη πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και το Ισραήλ έχει προσαρτήσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 67 και αυτό είναι αδιαπραγματεύσιμο. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Εάν οι Παλαιστίνοι δέχονται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με αυτή τη βάση είναι σαν να αυτοπυροβολούνται. Διότι Παλαιστίνοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί θα σημαίνει τότε παραδίδουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ στους Ισραηλινούς. Κανένας Άραβας ηγέτης δεν μπορεί ποτέ να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση. Τι σόι λοιπόν προσφορά κάνει ο Πρωθυπουργός τους Παλαιστίνιους όταν λέει αυτά. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε, ε, τελείως σε τέλμα. Σε τέλμα. Δεν υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία, δεν υπάρχει ειρηνευτική προσπάθεια, τα πάντα έχουν τελματωθεί. Θα με ρωτήσετε, με ποιο τρόπο θα βγούμε από αυτό το τέλμα. Και εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου λέω ότι η διέξοδος κατά τη γνώμη μου είναι μία και μόνοι. Οι μεγάλες δυνάμεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, Ρωσία να αποφασίσουν οι παράμετροι για μία συμφωνία θα οριστούν σε μία δήλωση που θα γίνει από το κουαρτέτο και θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και, και δεν λέω μία μια συμφωνία που θα επιβληθεί. κανένα δεν θέλει να του επιβληθεί μια συμφωνία. Αλλά εγώ λέω να καθίσουμε, να συμφωνήσουμε τις παραμέτρους, να συμφωνήσουμε ότι θα ιδρυθεί το Παλαιστινιακό κράτος, να συμφωνήσουμε ότι θα έχει μια ενιαία εδαφική κυριαρχία δεν θα χωριστεί σε καντόνια ώστε να μπορούν να το διασπάσουν οι Ισραηλινοί με αυτοκινητόδρομους α πούμε, που θα περνάνε μέσα από τι διάφορε. Ε, επαρχίες αν θέλετε, αλλά θα έχει μία ενιαία έκταση το Παλαιστινιακό κράτος αντίστοιχη με τις προστατευμένες περιοχές που τους ε, πήρε το Ισραήλ το 1967 και έτσι θα, και επίσης θα εξασφαλίσουν οι παράμετροι αυτοί την ασφάλεια του Ισραήλ στα εδάφη που είναι εντός των Ισραηλινών συνόρων και δεν θα υπάρχει καμία επέτηση για ε, Ισραηλινά εδάφη και παλαιστινιακά εδάφη τα οποία θα είναι εντός των συνόρων. Εάν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε αυτά, τότε οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι θα έλθουν να διπραγματευθούν με αυτές τις παραμέτρους τις οποίες θα τους βάλουμε στο τραπέζι. Θα πούμε ότι εσείς οι δύο δεν μπορείτε να τα βρείτε, άρα οι τέσσερις ε, εμείς σας θέτουμε αυτές τις παραμέτρους διαπραγμάτευσης και με αυτές θα καθίσετε στο τραπέζι. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ασφαλώς να αποτανθούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να αναζωογονήσει, να ανανύψει την ειρηνευτική διαδικασία. Ασφαλώς η Λιβύη, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, τους τελευταίους δέκα μέρες η Λιβύη προσπάθησε να εισαγαγεί ένα σχέδιο ψηφίσματος, παρουσίασε ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο ζητάει την αναστολή κάθε οικιστικής ενέργεια σε παλαιστινιακά εδάφη. Απλώς ζήτησε την αναστολή των ε, κατασκευαστικών διαδικασιών, την κατασκευή του χτισήματος δηλαδή, οικισμών, διότι ε, εάν συνεχιστεί αυτός ο κατασκευαστικός οριμαγδός δεν θα έχει μείνει και κανένα έδαφος για τους Παλαιστίνιους. Αλλά επειδή δεν βρήκαν ε, αρκετές ψήφους υποστήριξης, απέσυραν το ψήφισμα αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει ε, να γίνουμε σοβαροί. Εάν δεν μπορέσουμε με σοβαρότητα να σταματήσουμε την κατασκευή νέων οικισμούς, θα χαθεί κάθε ευκαιρία εδραίωσης, ε, εξασφάλισης των δύο αυτών κρατών. Έχουμε δύο λοιπόν εναλλακτικέ λύσεις μπροστά μας, όλοι, και εσείς και εμείς. Αφενός έχουμε τη σημερινή κατάσταση, δηλαδή ζητούμε μία διαπραγματευτική συμφωνία επί των παραμέτρων που σας ανέφερα ή δεν, μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουμε να τους πείσουμε Οπότε θα έχουμε άλλες δύο λύσεις, αν αποτύχουμε. Πρώτον, καταφυγή στη βία, ε, τρομοκρατία, χάος κοινωνικό και τα πολύ σιλιβερά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί επανειλημμένα στα τελευταία 15 χρόνια. Σκοτωμή, σαχισή αίμα, κάτι το οποίο βεβαίω με κάνει και να τριχιάσω. Αυτή θα είναι μία λύση αν αποτύχουμε και δεν είναι αποδεκτή από κανέναν. Δεύτερον, η, η άλλη αναπομένουσα λύση, εναλλακτική λύση, είναι χάος όχι μόνο για, τη, μια χώρα σαν τη δική μου, την Ιορδανία ε, και τις άλλες χώρες της ε, περιφέρειας, αλλά και χάος στην Ευρώπη. Διότι η Μεσόγειος είναι ε, δίπλα, βρέχει τα σύνορά σας. Οπότε, η μόνη λύση και η τελευταία λύση που παραμένει είναι μία χώρα με δύο λαούς. Θα δεχτεί ποτέ το Ισραήλ μία χώρα για δύο λαούς. Ποτέ. Ποτέ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να πιέσουμε τους Ισραηλινούς και να τους πούμε όχι, αποφασί, ε, αποφασίστε να σταματήσετε την οικιστική δραστηριότητα, ελάτε στο τραπέζι αρχίστε τις διαπραγματεύσει με τους Παλαιστίνους όχι επί τη βάση Ιουδαίας ε, και Σαμάρια, αλλά επί τη βάση της Δυτικής Όχθης. Όχι να. Εγώ δεν το, δεν το λέω αυτό η ειρηνευτική διαδικασία. Όταν ήμουν υφυπουργός, ε, το 1991 υφυπουργός ε, εξωτερικών στην Αίγυπτο, και ήμουν στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Γιτσακ Σαμίρ, είχε πει τότε το 81 ότι θέλουμε να, να ξεκινήσει ξανά η ειρηνευτική διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία και είχε πει, κοιτάξτε εγώ θα διαπραγματεύουμε με τους Παλαιστίνιους επί 10 χρόνια και θα τους δώσω μηδέν, μηδέν, στο τετράγωνο θα πάρουνε επί 10 χρόνια. Και τώρα τι βλέπουμε. Η κατάσταση επιδεινώνεται και αυξάνεται το, το, το κακό δηλαδή κάθε μέρα. Και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε, διότι όπως σας είπα η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι γειτονεύει και το Κοινοβούλιο με την αυξημένη νομοθετική του αρμοδιότητα, εξουσία, έχει τώρα περισσότερο από ποτέ τη δυνατότητα να παρέμβει, να κάνει κάτι ε, για αυτή την κατάσταση. Για τους Παλαιστίνιους τώρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να τους ενώσουμε. Έχουμε προτείνει κάποια συμφωνία, η οποία συμφωνία θα επέτρεπε στα δύο μέρη Αλφατάχ και Χαμάς να συνεργαστούν μέχρι ότου γίνουν οι εκλογές. Τη στιγμή που θα διεξαχθούν οι εκλογές, ο νικητής θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και θα προχωρήσουμε. Οι διαφορές μεταξύ Παλαιστινίων είναι επιζήμιες όσον αφορά τη δυνατότητα ειρήνευσης και επιζήμιες όσον αφορά την ενότητα του Παλαιστινιακού Εθνικού Κινήματος και εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Ισραήλ. Αν οι Παλαιστίνοι είναι διχασμένοι, νικούν οι Ισραηλινοί. Φυσικό είναι αυτό. Και το τίμημα δεν θα το πληρώσουν μόνο οι Παλαιστίνοι ή μόνο οι Ισραηλινοί. Όλοι μας θα το πληρώσουμε. Η Παλαιστινιακή Αρχή υπέγραψε τη συμφωνία που ετοιμάσαμε. Η Χαμάς αρνήθηκε να υπογράψει. Πρόβαλε κάποιες επιφυλάξεις, κάποια σχόλια. Σύντομα θα καταβληθεί εκ νέου Αιγυπτιακή προσπάθεια, ούτω ώστε να συμφωνήσουν. Ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουμε να τους πείσουμε να υπογράψουν μέχρι 24 Ιανουαρίου, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα, μέχρι 24 Ιανουαρίου κανένας, κανένας Παλαιστινιακός φορέας δεν είναι νόμιμος. Το Κοινοβούλιο θα είναι παράνομο, η Προεδρία θα είναι παράνομη και όλοι οι θεσμοί είναι άκυροι. Εκτός εάν σώσει την κατάσταση ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος. Πει θα εκδώσουμε προεδρικό διάταγμα αυτεξούσια σύμφωνα με το δίκαιο της Παλαιστίνης που θα ισχύει για όλους. Και θα καλύπτει τις εξουσίες τους μέχρι αυτή την ημερομηνία. Μέχρι να γίνει μάλλον να βρεθεί κάποια λύση. Είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια λύση. Νομίζω ότι μπορεί κάτι να συμβεί και όλοι θέλουμε να του υποστηρίξουμε να βρεθεί λύση, διότι εν τη ελλείψη ενότητος ε, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Αυτά όσον αφορά τις ενδοπαλαιστινιακές σχέσεις. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις όσον αφορά την ε, Ευρωμεσογειακή Ένωση. Η Ευρωμεσογειακή Ένωση, η Ένωση για τη Μεσόγειο μάλλον, δεν αποτελματώθηκε. Δεν έχει αποτελματωθεί η κατάσταση. Δεν έχει παγώσει, αλλά μία συνάντηση μόνο δεν πραγματοποιήθηκε. Μία σύνοδος υπουργών. Όλες οι άλλες συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα για το περιβάλλον, για το νερό, για τεχνολογία. Όλα αυτά λειτουργούν. Αυτό που αποτελματώθηκε ήταν η σύνθεση της γραμματείας όταν δεν έχει κανείς γενικό γραμματέα και γραμματεία δεν μπορεί να εφαρμόσει πράγματα ή να υλοποιεί προγράμματα. Και υπάρχουν έξι βασικά προγράμματα επί των οποίων θα πρέπει να εστιαστούμε. Στο Παρίσι την Κυριακή συναντήθηκα με το Γάλλο και Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών. Ισπανό διότι είναι η επερχόμενη Προεδρία Ισπανία και Γάλλο διότι είναι συνπροεδρός της πρωτοβουλίας η Γαλλία και αυτά που συζητήσαμε με κάνουν να πιστεύω και για την ώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Πιστεύω λοιπόν ότι σύντομα εντός εβδομάδων, το πολύ εβδομάδων, θα αρχίσει η λειτουργία της γραμματείας και θα συμφωνήσουμε πώς θα συνεδριάζει. Με τους ε, έξι αναπληρωτές γενικούς γραμματείς. Αυτά για την Ευρωμοσιακή Ένωση. Δεν νομίζω ότι οι σχέσεις Παλαιστινίων Ισραηλινών επηρεάζει την πρωτοβουλία. Γιατί το λέω αυτό. Διότι η πρωτοβουλία εδράζεται επί προγραμμάτων περισσότερο που εξυπηρετούν τη Μεσόγειο την Ευρώπη και τον Νότο και δεν εστιάζονται σε πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά ζητήματα θα βοηθούσαν αν επιληθούν. Να βρεθεί λύση. Αν έχουμε τη γραμματεία θα έχουμε και αναπληρωτή γενικό γραμματέα Παλαιστίνιο και Ισραηλινό αναπληρωτή γενικό γραμματέα. Όλοι αυτοί θα κάθονται γύρω από ένα τραπέζι κάθε πρωί. Θα συνεργάζονται με το γενικό γραμματέα και τους συναδέλφους τους. Θα προσπαθούν να διευκολύνουν τη λειτουργία της όλης πρωτοβουλίας. Ετέθηκε ένα ερώτημα για την Αίγυπτο και για την οικονομική κρίση, πώς επηρέασε την οικονομία μας. Η οικονομία μας μέχρι το 2008 ήταν στα 7,2-7,3% ποσοστό ε, ανάπτυξης ετησίως. Στόχος μας ήταν το 8% ετησίως μέχρι το 2009. Θεωρήσαμε ότι αυτό που μας περιόριζε και μας συγκρατούσε ήταν μόνο το πρόβλημα η έλλειψη σιδηροδρόμων και αυτοκινητοδρόμων. Αν είχαμε αρκετού σιδηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους, διότι βελτιώσαμε τα λιμάνια, αν τα βελτιώναμε σιδηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους για μεταφορά εμπορευμάτων, θα ήταν καλύτερα. Σιδηρόδρομοι και αυτοκινητόδρομοι μας περιόρισαν. Και ήμασταν πολύ φιλόδοξοι όσον αφορά αυτό το τομέα. Είχαμε ετοιμάσει σχέδιο, έρχεται η οικονομική κρίση και δυστυχώς πάμε στην ανάπτυξη 4,3, 4,4% φέτος. Κάποιοι θα έλεγαν, ωραία, 4,4, πολύ καλό είναι. Ναι, αλλά υπολογίστε και από πού ξεκίνησα, ε? από πού ξεκινήσαμε. Ελπίζαμε να είμαστε στο 8 με 9 και πέσαμε στο 4,4. Αυτά όσον αφορά την Αιγυπτιακή οικονομία ετέθηκε ένα ερώτημα όσον αφορά τους, τα τζαμιά και τους μιναρέδες στην Ελβετία. Λυπηρών. Θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι λαοί ο ένας τον άλλον στη Μεσόγειο. Γιατί το λέω αυτό. Βλέπετε τα τελευταία 10-15 χρόνια μιλάμε για διάλογο μεταξύ θρησκειών, μεταξύ πολιτισμών, διαπολιτισμικό διάλογο, διαθυσιστικό διάλογο, συμμαχία πολιτισμών όσον αφορά την Ισπανία και την Τουρκία. Παρουσιάστηκαν ιδέες από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, παρέστημεν σε συζητήσεις στην Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας και στο Ίδρυμα Άννα Λίντ, που εκεί συζητήθηκε το θέμα και ξαφνικά Όλα αυτά τα ρίχνουν πίσω. Τα πετάνε στα μούτρα της μουσουλμανικής κοινότητας της Ελβετίας. Και βλέπω ότι κάποιοι σε ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να συμβουλεύσουν παρόμοια προσέγγιση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια θλιβερή εξέλιξη και αυτό είναι το λιγότερο που έχω να πω. Θα δείξει ότι κάποιες κοινωνίες δεν είναι αρκετά ανοιχτέ. Και όχι μόνο αυτό, κάποιες ε, κοινωνίες δίνουν σύμβουλες, μιλάνε για κάποια θέματα, λόγια μεν, διαφορετικά τα οποία δεν εφαρμόζονται στις κοινωνίες τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό είναι το λιγότερο μπορεί να πει κανείς. Πώς επηρεάζει αυτό τους Αιγυπτίους κόπτες, έτσι επηρεάζει καθόλου. Όποιος επισκεφτεί την Αίγυπτο, ή επισκέπτεται την Αίγυπτο, βλέπει εκκλησίες παντού και δεν θεωρούμε την κοπτική κοινότητα της Αιγύπτου μειονότητα. Διότι συχνά μειονότητες είναι διαφορετικής εθνότητας. Οι κόπτες είναι Αιγύπτιοι συχνά αποκαλούνται ή αυτοαποκαλούνται πιο Αιγύπτιοι από τους υπόλοιπους. Διότι πάντα ήταν εκεί. Τίποτα δεν τους επηρεάζει, είναι Αιγύπτιοι. Τους υπερασπιζόμαστε, τους στρατολογούμε, τους προσλαμβάνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, προσλαμβάνονται και διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κοινότητα. Τώρα, σχέσεις Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προώθησης βελτίωσης αυτών, το επεξεργαζόμαστε. Υπάρχει μια επιτροπή. Ήταν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα προετοιμάζει και θα εξετάζει τρόπους ε, βελτιώσεως αναβαθμίσεως των σχέσεων των δύο μέρων και θα γίνει συνεδρίαση Συμβουλίου Σύνδεσης περίπου Απρίλιο, 26-27 Απριλίου. Εκεί θα δούμε ποια είναι η πρόοδος που επετεύχθη. Ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για μια χώρα όπως είναι η Αίγυπτος ο μεγαλύτερος εταίρος μας ο εμπορικός είναι η Ευρώπη. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται τη σημασία της Αιγύπτου από όλους. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω. Δηλαδή, η Αίγυπτος ανήκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα πριν πολύ Ευρωπαίοι μπήκαν να μπουν στην αυτοκρατορία. Είχαμε συναλλαγές με την Ελλάδα, με τη Ρώμη, με την Ισπανία, με την Κύπρο, με τη Μάλτα. Πολλές λέξεις μας έχουν ρίζες ελληνικές ή ιταλικές. Οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή μεταξύ Αιγύπτου και μελών μεσογειακών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σχέσεις ε, που δεν έχουν όριο. Υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες ε, βελτιώσεως των σχέσεων. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που ετέθη για το Αφγανιστάν. Πολύ δύσκολο να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Όμως πρέπει να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Το θέμα του Αφγανιστάν δεν θα ρυθμιστεί με τη χρήση βίας. Η βία ισχύς είναι μόνο μία συνιστόσα. Όμως πρέπει να εστιάζεται επί πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών μέσων. Επιλέγει στατιωτική επιλογή και τότε κολλάς αιωνίως αν την επιλέξεις, αιώνια. Και η βία θα αυξάνεται. Και ο Αφγανός δεν υποκύπτει με τη βία, διότι βλέπει τον ξένο και τον θεωρεί εχθρό του. Και από τη στιγμή που υπάρχει ξένος στη γη του, σε αυτή την άγωνη γη του θα πολεμάει. Να είσαστε σίγουροι θα πολεμάει. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι αν θέλετε να αυξήσετε την παρουσία δυνάμεων, τότε τις αυξάνετε για πολύ σύντομη χρονική περίοδο, μέχρι τη στιγμή που δημιουργείται ντόπια αυγανική δύναμη που θα ελέγχει την κατάσταση στη χώρα. Και όχι σε όλη τη χώρα. Διότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του βασιλείου ή της δημοκρατίας πριν την παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης, το Αφγανιστάν ήταν μια χώρα που ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Οπότε γίνεται κάποια συνεννόηση με τις διάφορες δυνάμεις, με τις διάφορες δυνάμεις, τις επιτόπιες. Λέω διάφορες δυνάμεις, όλες εννοώ τις επιτόπιες δυνάμεις. Εγώ μετά προσπαθείς να οικοδομήσεις την οικονομία της χώρας, μετά προσπαθείς να χρηματοδοτήσεις τα στοιχεία, να πιέσεις μάλλον, να στριμώξεις τις δυνάμεις που συνθλίβουν την κεντρική εξουσία και ελέγχεις επίσης και το εμπόριο ναρκωτικών. Το εμπόριο ναρκωτικών βοηθά κάποια στοιχεία της κοινωνίας που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Οικονομικά στοιχεία, πολιτικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία, μέσα μάλλον, συγγνώμη, στατιωτικά μέσα, δεν θα κάνουν τη δουλειά, δεν θα βρουν λύση. Είναι μια μουσουλμανική κοινωνία. Προσέξτε το αυτό. Διότι κάθε φόνος μουσουλμάνου στο Αφγανιστάν γίνεται αισθητό στο Μαρόκο. Ο πυροβολισμός, ότι η τυφλή χρήση όπλων που σκοτώνει κάποιον ηγέτη και ταυτόχρονα όπως προσπαθεί να σκοτώσει τον ηγέτη, σκοτώνει και 10 οικογένειες, είναι κάτι που σε κυνηγάει, κυνηγάει εσένα και τα στατεύματά σου. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Είχαμε εμπειρία τέτοιων γεγονότων το 62 με 68 στην Ιεμένη. Πολύ δύσκολη εμπειρία, λόγω εδάφους, λόγω φυλών, λόγω εθνοτήτων. Είναι μια κοινωνία που πρέπει να την καταλάβεις πριν ξεκινήσεις για να κάνεις κάτι. Έχουμε τρία ερωτήματα που απομένουν. Σαλίντ, ο Ιζαρινός στρατιώτης Σαλίντ. Επεξεργαζόμαστε ένα πακέτο. Οι Ισραηλινοί θα πρέπει να δεσμευτούν. Αποφάσισαν οι Ισραηλινοί να δεχθούν, να πληρώσουν χρήματα για τον Σαλίντ. Τίμημα χίλιους Παλαιστίνιους σαν τάλαμα για αυτόν από τους 12 φυλακισμένους. 12.000. Κανείς δεν ξέρει τα ονόματα των 12.000 κρατουμένων Παλαιστινίων. Όσο και να σκέφτεται κανείς ένα στατιώτη, είναι μια ζωή, το δέχομαι, υπερασπίζομαι στο και μια ζωή, αλλά έχω 12.000 Παλαιστινίους σε Ισραηλινές φυλακές. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός. όσο και αν μας νοιάζει, ε, ε, αυτό είναι θέμα διοντολογίας επί αρχών. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Οι Ζαλινοί κάνουν ένα βήμα προς τα μπρος, δύο προς τα πίσω. Τι λέω, τι εννοώ. Δηλαδή, δέχονται να απελευθερώσουν χίλιους κρατουμένους, αλλά παζαρεύουν τα ονόματα. Ποιους θα απελευθερώσουν. Αυτός έχει αίμα στα χέρια του. Ο άλλος έχει κάνει κάτι άλλο, έχει άλλο στα χέρια του. Δεν είναι αυτή η λύση. Ποια είναι η λύση. Λέμε, καλώς, Ζητάς χίλιους. Δώσ' μου τα ονόματα, θα σου δώσω τους χίλιους. Τελεία και παύλα. Διότι στο κάτω-κάτω θα ζουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και αν αποφασίσεις να τους ξαναμαζέψεις σε μια νύχτα, ξανά τους ξαναμαζεύεις. Εν μια νυχτή. Γιατί να κολλήσει εργής, γιατί να παίζει παιχνίδια. Αυτά για τον Σαλίτ. Τώρα, για αυτό που αποκαλείται... Ξέρω τι να σας πω για το Ιράν. Οι Ισραηλινοί σταμάτησαν ένα-δύο πλοία στην ανοιχτή θάλασσα, στη Μεσόγειο. Τα πήραν τα πλοία στη Χάιφα. Εκένωσαν κάποιο εμπόρευμα που ίσως, ίσως, ίσως και όχι, να ήταν ύποπτο. Δεν υπήρχαν ανεξάρτητοι παρατηρητές. Αν τέτοια φορτία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ, εμείς θα έχουμε αντιρρήσει έναν αντιχώρο που θέλει να χρησιμοποιήσει τη διόρυγα του Σουέζ για να στέλνει υλικό παράνομο ή που δεν ανταποκρίνεται στο, στη φορτω, φορτωτική του πλοίου. Διότι όταν λέει ότι μεταφέρει ε, σιτάρι το πλοίο στη φορτωτική, θα πρέπει πράγματι να περιέχει σιτάρι και όχι πυράβλος κατιούσα. Όμως ε, αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας να μπορούμε να βλέπουμε ακόμα τι γίνεται και μέσα στα εμπορευματοκιβώτια. Αλλά δεν μπορείς να... να μαζεύουμε εμείς τα πλοία και να τα φέρουμε στα λιμάνια μας και να κατεβάζουμε εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια για να διεξαγάγουμε ελέγχους, αυτό είναι πάρα πολύ δαπανήρο. Καθυστερήσεις δημιουργεί. Και τα λιμάνια μας θα τα αποφεύγουν. Θα αποφεύγει ο κόσμος να έρχεται στα λιμάνια μας αν το κάνουμε αυτό. Αλλά θα είναι και παχθής διαδικασία αν το ακολουθήσουμε αυτό. Η άποψή μας όσον αφορά τις νέες δυνατότητες, τις νέες μονάδες για εμπλουτισμό, τις 10 όπως εικάζεται, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που εκνευρίζει τους Ιρανούς αδελφούς μας. Είναι θυμωμένοι οι Ιρανοί αδελφοί μας και ίσως λένε πράγματα τα οποία δεν θα κάνουν τελικά και δεν χρειάζεται να τα κάνουν. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται 10 μονάδες εμπλουτισμού. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και σας παρακαλώ να με ανεχθείτε σε αυτό που λέω, να με καταλάβετε αυτό που πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να επιμείνουμε είναι στο δικαίωμα των χωρών να χρησιμοποιούν με ειρηνικό τρόπο την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικού σκοπούς. Οι χώρες πρέπει να δρουν με τρόπο τέτοιο που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη, που θα μεταδίδει ε, εμπιστοσύνη. Αλλά το δικαίωμα κάθε χώρας για την ειρηνική χρήση της πυρηνική ενέργεια σύμφωνα με ε, την συνθήκη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια. Εάν μια χώρα συλληφθεί να κάνει παράνομα πράγματα και είναι μέλος του καθεστώτος αυτού, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να την εντοπίσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πρέπει εκεί στην περιοχή μας να έχουμε μια περιοχή, μια ζώνη που θα είναι ελεύθερη από πυρηνικά όπλα. Υπάρχει μια χώρα στην περιοχή, το Ισραήλ, που δεν είναι μέλος του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και καλούμε το Ισραήλ να προσχωρήσει στο σύμφωνο αυτό μη διάδοση των πυρηνικών όπλων αλλά να δεχθεί επίσης και τη δημιουργία μιας τέτοια ζώνης που θα είναι ελεύθερη από πυρηνικά όπλα. Δεν το κάνει κανείς αυτό δεν ακολουθεί κανείς αυτή τη δια... αν δεν κάνει κανείς αυτή τη διαδικασία, τότε τίθεται εν κινδύνο όλη η Μεσόγειος. Όλη η Μεσόγειος. Μην θεωρείτε ότι η Ελλάδα ή η Κύπρος δεν θα επηρεαστούν. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να, προκύρι να δημιουργηθεί μια ζώνη τέτοια και να πάμε στους Ισραηλινούς και στους Ιρανούς και να τους πούμε ακούστε εδώ αυτό θέλει η διεθνής κοινότητα και οι δυο σας Ισραήλ από τη μια πρέπει να παραιτηθείτε από τη δυνατότητα των πυρηνικών όπλων και το Ιράν πρέπει να δώσει διαβεβαιώσει στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν έχει σαν στόχο την απόκτηση πυρηνικών όπλων.